<clears throat> Good morning. Good morning. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην τρίτη ενότητα της κοινή μα συνεδρίασης. Με μεγάλη τιμή καλώς ορίζω την κυρία Βάλστρομ, βασική μας ομιλήτρια για σήμερα, τον Μάικλ Κάσμαν, τον κύριο Μάικλ Κάσμαν και ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του συναδέλφου Αλεξάνδρου Βόντρα που είναι γερουσιαστής και αντιπρόεδρος της τσεχικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε βοτιλιάρισμα μεταξύ αεροδρομίου και εθούσης κάπου. Θέλω να θυμίσω τη συνθήκη και συγκεκριμένα το πρώτο άρθρο και το δεύτερο που ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει όσο γίνεται με μεγαλύτερη διαφάνεια αποφάσεις και όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Το άρθρο 253 λέγει ότι Όλοι οι πολίτες και διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δικαίωμα πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα έγγραφα μάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες στο άρθρο 42 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Βεβαίως με κανόνες που και εξαιρέσεις που ορίζονται λεπτόμερος στον ε, εκτελεστικό κανονισμό 1049 του 2001. Τον Απρίλιο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση για εφαρμογή και κάποια κράτη ε, το θεώρησαν αυτό που στο στη διαφάνεια. Η σημερινή μας συνεδρίαση αποτελεί καλή ευκαιρία ε, συζήτησης αυτής της πρότασης. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τον συνάδελφο Μάικλ Κάσμα να λάβει το λόγο. Thank you uh, good morning, everyone. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους. Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω ε, στην ενότητα που ε, είναι αφιερωμένη στην πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Εργαζόμενος σε αυτόν τον κανονισμό, αισθάνομαι ως δύο χαρακτήρες του Σέξπι, τον Πρόσπερο στη Θίελα που ε, είναι ονειροπόλες και το Μαλβόλιο ε, από άλλο θεατρικό ε, που τελικά έχει κακό τέλος. Ελπίζω να είμαι ο, ο πρόσπερος, ο πρώτος χαρακτήρας, το πράγμα που επιθυμούν και πολλοί πολίτες της Ένωσης και πολλοί που απευθύνονται σε εμά. Όπως είπε ο Πρόεδρος, εδώ πρόκειται για ένα θεμελιώδες δικαίωμα και η πρόσβαση στα έγγραφα, η πρόσβαση στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση είναι το μέσον εκείνο με το οποίο Μπορούν οι πολίτες, ε, άτομα, ε, ατομικά αλλά και συλλογικά να μας ε, φέρουν ενώπιον των ευθυνών μας και να είμαστε υπόλογοι στα μάτια τους. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το τι κάνουμε, αλλά το τι κάνουμε και πώς αυτό παρουσιάζεται και παρερμηνεύεται ή διαστρεβλώνεται. Έτσι λοιπόν η πρόσβαση στο στα έγγραφα και στην ενημέρωση είναι ζωτική σημασία. Αν θέλουμε οι πολίτες να καταλάβουν τι κάνουμε. Αν δουν οι πολίτες τους υπουργούς τους να ψηφίζουν και να συζητούν δημόσια στο Συμβούλιο, θα καταλάβουν ότι θα είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν οι υπουργοί επιστρέφοντα στα κοινοβούλια του και να μην τα ρίχνουν όλε τι Βρυξέλλε εντό εισαγωγικών. Γιατί θα έχουν δει οι πολίτε πώ λαμβάνουν οι αποφάσει και σε ποιε συζητήσει στο Συμβούλιο και με ποιε ψηφοφορίε. Όταν λοιπόν προετοιμάσαμε το 1999 τον κανονισμό αυτό μέχρι το 2001 και χαίρομαι που παρευρίσκεται η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Βάλστρομ γιατί συμμετείχε και εκείνη τότε στην αρχική ακόμα φάση όταν λοιπόν ξεκινήσαμε διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα κενό που έπρεπε να πληρωθεί. Πριν από αυτό, το δικαίωμα του κοινού στην πρόσβαση και στα έγγραφα δεν ήταν δικαίωμα, ήταν ένα δώρο που έκαναν τα θεσμικά όργανα στους πολίτες τους πρόσφερα αυτή τη δυνατότητα. Και εμείς θελήσαμε να κατοχυρωθεί ε, ως αρχή η πρόσβαση στα έγγραφα και η εξαίρεση να είναι η απαγόρευση κατά περίπτωση κάθε φορά. Αναθεωρώντας λοιπόν το έγγραφο και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εξετάζοντας, δουλεύουμε με την εμπειρία του 2001 αλλά και με βάση την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και χαίρομαι που βλέπω εδώ τον κύριο Τούρκο και τον καλωσορίζω, ο οποίος ήταν πραγματικά πρωταγωνιστής στην αναθεώρηση ε, της πρότασης αυτής. Εκείνοι από εσάς που θα έχετε ίσως δει την έκθεσή μου ή το σχέδιο έκθεσης, διαπιστώσατε ότι καλωσορίζω την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής με κάποιες επιφυλάξεις μεν, ε, αλλά λέω ε, και ξεκάθαρα ότι δεν είναι παρκής στη φιλοδοξία της. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που δικαιολογούνται, όπως είναι ε, η διεύρυνση των δικαιούχων και ε, ο συντονισμός ε, της πρότασης αυτής με τη σύμβαση του Άρχους. Βέβαια υπάρχει και οπισθοδρόμηση. Το 2006 είχα συντάξει ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε τελικά από το Κοινοβούλιο, αλλά τα περισσότερα από όσα λέμε εκεί δεν ελήφθησαν υπόψη. Θα ήθελα επί ευκαιρία να σας ε, αναφέρω ότι θέλω ε, τα θεσμικά όργανα να μπορούν να συνεργάζονται, να υπάρχει μια ιεράρχηση για κοινού κανόνε και κατευθυντήριε γραμμέ για να μπορούν να ανταποκρίνονται ε, στα διάφορα έγγραφα που είναι πολύ διαφορετικά τα ίδια εγγράφων. Ξέρετε ότι δεν ξεκινούμε από μηδενική βάση, διότι ήδη υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες. Ε, σε βάση υπείου δικαίου, όχι νομοθεσία, αλλά soft law. Και θέλουμε όλα, θα προσπαθήσουμε όλα τα θεσμικά όργανα να έχουν το ίδιο στόχο. βεβαίω ε, έχουμε διάφορα ε, συστήματα πληροφορικής, ε, ε, την υπηρεσία δημοσιεύσεων, την κωδικοποίηση που γίνεται σε κοινή προσπάθεια και την νομοπαρασκευαστική δουλειά. Θέλουμε οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων να καταστούν πιο Κατανοητέ. Θα ήθελα να πω στους παρόντες εθνικούς βουλευτές όταν αναφέρομαι στην ευρωπαϊκή λήψη αποφάσεων, η διαδικασία λήψη αποφάσεων δεν αφορά αυτό μόνο την Ευρώπη αλλά και ε, τις εφαρμοστικέ διατάξεις και μέτρα στα κράτη-μέλη γιατί αυτά τελικά είναι τα κείμενα που αφορούν και τους δικού σα πολίτε και τους ε, δικού μα. Εκείνη που με γνωρίζετε δεν θα εκπλαγείτε. Η δική μου πρόταση είναι πολύ πιο φιλόδοξη από εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμα και μεγαλύτερη από την προθυμία του Συμβουλίου. Εγώ προσπαθώ να οικοδομήσω στην κοινή μας εμπειρία ε, από τη θεσμική σκοπιά θα πρέπει να συμμεριζόμαστε όλοι τα καθήκοντα και τους στόχους και τους σκοπούς μας σύμφωνα με τις συνθήκες. Και υπό την έννοια αυτή προσπαθώ να καλύψω το έλλειμμα ε, κοινών κανόνων για τα διαβαθμισμένα έγγραφα. Υπάρχουν μερικοί που θεωρούν ότι όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι δημόσια, χωρίς καμία διαβάθμιση. Και κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ε, προσβάσιμα στο κοινό. Αυτό βέβαια είναι τελείως αναφάρμοστο στην πράξη. Αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει καμία διαβάθμιση των εγγράφων και καμία εμπιστευτικότητα, τότε τα θεσμικά όργανα σίγουρα σε σχέση με τους διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς θα ε, ε, αντιδράσουν. Εγώ προσπαθώ να πετύχω τον υψηλότερο στόχο, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και τα θεσμικά όργανα και οι θεσμοί και οι βουλευτές θα πρέπει κάπου να ε, έχουν και εξαιρέσει και ε, ε, εμπιστευτικά έγγραφα. Εκείνοι που γνωρίζουν το κανονισμό ε, ξέρουν ότι υπάρχει το άρθρο 9 που ορίζει τα λεγόμενα ευαίσθητα έγγραφα και ασχολείται με αυτό το θέμα της διαβάθμισης των έγγραφων. Θα ήθελα να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό το θέμα και με τις καλές αρχές που έχει το Συμβούλιο στον ιστορικό κανονισμό του αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. στο βαθμό που μπορούν αυτά όμως να μεταφερθούν ως αρχές σε ένα κοινοβουλευτικό σώμα. Δεύτερη πρόκληση. Θα πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε, ε, στη διαφάνεια, τη νομοθετική και τη διοικητική διαφάνεια. Ευκαιρία, εξήγησα ποια είναι η διαφανής και καλή διοίκηση ε, στο άρθρο 41 άλλωστε του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, ορίζονται όλα αυτά. Επειδή τελειώνει ο χρόνος μου, Πρόεδρε, θα ήθελα ε, συμπεραίνοντας να σας συστήσω να διαβάσετε την αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο έκθεσής μου. Θα δείτε ότι αναφέρομαι σε κάποιες τροπολογίες και μεταξύ αυτών ο διαχωρισμός του πεδίου εφαρμογή τη οδηγία από τους δικαιούχου. Επίσης, για τους ορισμούς αποφάσισα να επαναφέρουμε ε, τον παλιό ορισμό του εγγράφου, TST έγγραφο, όπω ορίζεται από το σημερινό κανονισμό, γιατί είναι πολύ ευρύτερη και πλήρης και θα πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο και ιστορικά έγγραφα, ε, νομοθετικού περιεχομένου και διοικητικά έγγραφα. Ε, στις εξαιρέσεις να γίνεται διάκριση μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, καθεστώς με βάση το οποίο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει έγγραφα τρίτων μερών, που μέχρι τώρα αυτό προκάλεσε πολλά προγράμματα ε, στη θεσμική καθημερινότητα. Επίσης, μιλώ ε, καλημέρα σας και καλώς ορίστε κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, για το ρόλο και την ευθύνη της ενημέρωση, του, του υπαλλήλου που οφείλει να ενημερώνει στην υπηρεσία δημοσιεύσεων. Να είναι υπεύθυνος για το πρωτόκολλο, για το αρχείο και ε, να ε, βεβαιούται ότι κάθε γενική διεύθυνση ε, συμμορφούνται προς τις υποχρεώσεις της και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Ο ρόλος και ευθύνη του υπαλλήλου αυτού είναι πρωταγωνιστικός επίση πιστεύω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε το ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που να αποτελεί σημείο αναφορά στα θεσμικά όργανα για του υπευθύνου τη πληροφόρηση και να ε, προσφεύγουμε στο Διαμεσολαβητή ε, όταν υπάρχει κάποια αμφιβολία. Και ε, αναφέρομαι επίση τέλο σε μια τροπολογία για τι κυρώσει σε περίπτωση που μια χώρα δεν συμμορφώνεται. Θέλω να τελειώσω όπω ξεκίνησα. Μερικοί θα πούν ότι είμαστε φιλόδοξοι, Α, ότι δεν πρόκειται να καταφέρουμε το στόχο μας αυτό. Θυμάστε τι το Σάντσο Πάντσα. που έλεγε ποτέ δεν θα σπάσεις τη λόγη σου αν δεν ε, επιτεθείς σαν Σε ευχαριστώ πολύ. Thank you very much for your speech. Ευχαριστούμε πολύ για την εισήγηση αυτή κύριε Μιχαήλ Κάσμαν. Καλωσορίζω τον Αντιπρόεδρο της ε, τσεχικής δημοκρατίας και του δίνω το λόγο. Α, ναι, εντάξει. Ευχαριστώ Ρούντεκ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα αλλά υπήρχε κακοκαιρία και πολύ μεγάλη κυκλοφορία στις Βρυξέλλες. Βλέπω ότι γνωρίζω πολλούς εδώ Καταρχήν ευχαριστώ τους οργανωτές της κοινή αυτής συνεδρίασης για την πρόσκληση που μου έκαναν να περιγράψω τις ζωτικές πτυχές της πρότασης της Κομισιόν για την αναθεώρηση του κανονισμού 1049 για την δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσιμών. Δεν ξέρω αν το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια πρόσεξαν δεόντως το θέμα αυτό. Εγώ είμαι μέλος και της Τσεχικής Γερουσίας και γνωρίζω ότι ο Λούμπολ Τσέφτσικ και άλλοι το προσέχουν ιδιαίτερος. Ίσως ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Απρίλιο υπέβαλε την πρότασή της για αναθεώρηση του προηγούμενου κανονισμού για την πρόσβαση στα έγγραφα και την υπέβαλε αυτήν την πρόταση κανονισμού με τη μορφή αναθεωρημένης πρότασης. Η Προεδρία δέχεται την επιλογή αυτή. Θεωρεί πολύ σημαντικό οι κανόνες που εφαρμόζονται για αυτό το θέμα να είναι σαφείς και, και ευνόητοι. Η επιλογή αυτή του recasting που λέμε ε, σημαίνει ότι η τεχνική αυτή στοχεύει στην διευκόλυνση της πρόσβασης στις αλλαγές και αναθεωρήσεις των νομοθετικών κειμένων. Τώρα για τα πρακτικά. Το Συμβούλιο βέβαια γνωρίζει ότι χρειάζεται ενημέρωση του κανονισμού 1049 αλλά παραμένει πεπισμένο ότι ο κανονισμός αυτός γενικά έχει λειτουργήσει πολύ καλά. Από τότε που τέθηκε ενισχύ το Δεκέμβριο 2001, το Συμβούλιο και ο Γενικός του Γραμματεύς έλαβαν πολλά μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη και σωστή εφαρμογή των κανόνων διαφανείας. Ένα από αυτά τα μέτρα ήταν να δημιουργηθεί ένα κεντρικό μητρό ενιαίο ακόμη πριν, πριν ακόμα αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός αυτός. Ήδη τον Ιανουάριο ε, του 89 γινόταν αναφορά σε ανώτατο όριο χιλίων εγγράφων. Και αυτό θεωρήθηκε τελικά συμβουλιακό έγγραφο και όχι έγγραφο από την Κομισιόν ή από άλλες πλευρές. Έτσι στις συζητήσεις του Συμβουλίου και των επιτροπών του και των ομάδων εργασίας του οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των χωρών μελών δεν είναι πρόσωπα ή οντότητες εκτός των θεσμών αλλά ανήκουν σε αυτούς. Η αρχή αυτή βοήθησε το Συμβούλιο και τη Γενική του Γραμματεία να διεκπαιρεώσουν πολλά αιτήματα για πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τη δουλειά του Συμβουλίου και των προπαρασκευαστικών του σωμάτων με αποτελεσματικό τρόπο. Όσο για την πρόταση τώρα της Κομισιόν που εξετάστηκε από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την πληροφόρηση, ας σας πω τα εξής. Η εξέταση της πρότασης της Κομισιόν από την ομάδα εργασίας πληροφόρησης του Συμβουλίου στο δεύτερο μισό του 2008 βασικά ήταν τεχνικού χαρακτήρα και μπορεί κανείς να κάνει μερικές γενικές παρατηρήσεις από αυτήν την διεκπαιρέωση. Πρώτον, για το άρθρο 2 για τους δικαιούχους ή αυτούς που ωφελούνται από αυτές τις διαδικασίες αποκλείεται εκεί η δυνατότητα επέκτασης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του κανόνα αυτού ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικία στην εθνικότητα του ετούντος. Αλλά σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος κανονισμού τα θεσμικά όργανα μπορούν να δώσουν πρόσβαση σε πρόσωπα που δεν παραμένουν ή δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κάποια ενωσιακή χώρα. Δεν εμποδίζει τίποτα το θεσμικό όργανο να δώσει, να χορηγήσει πρόσβαση και στο μέλλον αλλά σύμφωνα με τον εσωτερικό του κανονισμό του κάθε όργανο. Το άρθρο 3 που είναι ο ορισμός του TST έγγραφο θεωρεί ως έγγραφο τα δεδομένα που έχουν τη διατηρηθεί σε ηλεκτρονικές τράπεζες δεδομένων εφόσον μπορούν να τυπωθούν ή να σταλούν με τυπώσιμη μορφή. Το 4.1 και το 4.4 μιλούν για την εφαρμογή του κανονισμού του άρχους, του κανόνα του άρχους, όπου γίνεται λόγος για την ευθυγράμμιση της πρόσβασης με αυτά που προβλέπονται για τις πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον στον κανονισμό 1367 του 2006 Εκείνο τον κανονισμό που τον λέμε κανονισμό του άρχους ο, μετά το, τα άρθρα 4 και 5 δηλαδή η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα εδώ το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στην περίπτωση Λάγκερ εξετάζει ακόμη την υπόθεση σε έφεση και γι' αυτό μέχρι το βγει απόφαση παραμένουν οι ισχύουσες διατάξεις διότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα βγάλει τελικά την απόφαση σε μερικούς μήνες. Το Συμβούλιο λοιπόν περιμένει το αποτέλεσμα της εξέτασης της ε, πρότασης αναθεώρησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή σας ευχαριστώ λοιπόν. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης και Αντιπρωθυπουργέ. Και τώρα το λόγο έχει ο επόμενος ομιλητής, δηλαδή η κυρία Βάλστρομ, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνη για τις ε, σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, εξοχότατοι και εξοχότατες. Το δικαίωμα στη γνώση και πληροφόρηση είναι σημαντικό για τη δημοκρατία, όσο και το δικαίωμα ψήφου. Και για να υπάρχει χρειάζεται, χρειάζονται κατάλληλα εργαλεία, διαφάνεια και δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα. Από εκεί πρέπει να αρχίσουμε σε ποιες αρχές πρέπει να βασιστούμε και ποιος είναι ο τελικός μας στόχος. Αφού συμφωνήσουμε αυτά μπορούμε να συζητήσουμε τους τρόπους, τα μέσα για να τα πετύχουμε. Τεχνικά μέσα και διαδικασίες. Κατά τα λίγα λεπτά που διαθέτω θα ήθελα να σας αναφέρω τέσσερα κύρια σημεία. Πρώτον, ο κανονισμός 1049 λειτουργήσε καλά τα πρώτα 7 χρόνια της εφαρμογής του δεν χρειάζονται τεράστιες αλλαγές αλλά μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις. Δεύτερον, οι επαγγελματίες στα ευρωπαϊκά χρησιμοποίησαν επανειλημμένως τον κανονισμό και τώρα πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση και για τους απλούς πολίτες. Τρίτον, η πρόταση της Κομισιόν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη και όχι λιγότερη διαφάνεια. Οποιοδήποτε έγγραφο που μπορεί να χορηγηθεί με τους ισχύοντες κανόνες θα μπορεί να χορηγηθεί και με τους αναθεωρημένους. Και τέταρτον, δεν χρειάζονται τεράστιες αλλαγές, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μητρώα και τις ιστοσελίδες. Εκτός από αυτά τα τέσσερα σημεία θα προσπαθήσω να σχολιάσω και ορισμένα στοιχεία που ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής. Δεν υπήρχαν previous speakers, μόνο ένας έτσι ώστε να υπάρξει στη συνέχεια μια συζήτηση και η μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της γνώσης των εθνικών βουλευτών. Από το 1992 οπότε και νεκρήθη η δήλωση για το δικαίωμα στην πρόσβαση στα έγγραφα έχουν αλλάξει μερικά πράγματα. Από τότε όμως ήδη είχε διατυπωθεί η πρώτη αρχή. Η διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων είναι βασική για το δημοκρατικό χαρακτήρα της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων και για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και διοίκησης. Σε αυτά βασίστηκε λοιπόν το 2001 ο κανονισμός 1049 και αυτή η αρχή συνεχίζει να διέπει και την αναθεώρησή του για το μέλλον. Εφτά χρόνια εμπειρίας λοιπόν της λειτουργίας του κανονισμού αυτού προκάλεσαν την ανάγκη για ορισμένες αλλαγές, βελτιώσεις. Υπήρξε μεγάλη αύξηση των ετοιμάτων για πρόσβαση και όλο και λιγότερες αρνήσεις. Από την άλλη μεριά όλο και περισσότερες πληροφορίες χορηγήθηκαν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στην πράξη. Έτσι λοιπόν χρειάζεται, καταλάβαμε ότι χρειάζεται μία πιο ενεργή στάση για την ενημέρωση του ισχύοντος κανονισμού. Επίσης είδαμε ότι ο κανονισμός συνήθως χρησιμοποιείται από εταιρείε νομικά γραφεία και λομπιίστες. Δεν το χρησιμοποιούν τα θέματα που ενδιαφέρουν όλους αυτούς δεν είναι μόνο η νομοθεσία αλλά κυρίως η εφαρμογή της, ο τρόπος εφαρμογής της. Δεν μπορώ να πω ότι ωφελήθηκε και πολύ ο απλός πολίτης, ούτε καν η δημοσιογράφη. Τα τελευταία δύο χρόνια αρχίζει να υπάρχει μεγαλύτερη χρησιμοποίησή του από τον ακαδημαϊκό κόσμο. Ο γενικότερος στόχος της Κομισιόν για την αναθεώρηση του κανονισμού είναι πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τη λήψη αποφάσεων να δοθεί στο, σε ευρύτερο κοινό. Να υπάρχει πιο ενεργή διάδοση των εγγράφων και να ευθυγραμμιστεί το 1049 με τις διατάξεις που οδηγούν στη δημιουργία του ενιαίου πλαισίου για τη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα καθώς και τη σύνδεση του 1049 με άλλα νομικά εργαλεία που αφορούν και αυτά την πρόσβαση στα έγγραφα. Ορισμένα τμήματα της πρότασης της Κομισιόν έχουν θεωρηθεί σαν υπαναχωρήσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι αντικειμενικά λάθος, αλλά δείχνει ότι δεν τα είπαμε και πολύ καθαρά. Ας προσπαθήσω να διορθώσω τα πράγματα λοιπόν. Τέσσερα θέματα έχουν γίνει αντικείμενο επικρίσεων. Πρώτον, ο προτινόμενος ορισμός του TST έγγραφων. Δεύτερον, η εξισορρόπηση μεταξύ χορήγησης πληροφόρησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τρίτον, το δικαίωμα των κρατών μελών να αντιταχθούν στην διάδοση πληροφοριών που έχουν χορηγήσει στα θεσμικά όργανα και τέταρτον η απαγόρευση της πρόσβασης υπό ορισμένε εξαιρέσεις. Το περίφημο άρθρο που αφορά αυτές τις προσωρινές εξαιρέσεις. Πρώτον λοιπόν, ο ορισμός του εγγράφου. Εδώ προτείναμε αλλαγή διότι ο ισχύων ορισμός δεν είναι ακριβής αφήνει χώρο για αυθαιρεσίες, αυθαίρετες ερμηνείες. Εμείς θέλουμε ο να είναι σαφέστερος και γι' αυτό κάνουμε δύο αποσαφηνείς των ισχύοντα. Ένα έγγραφο που γράφεται επισήμως από κάποιο όργανο έχει, έχει υποβληθεί στον δικαιούχο ή έχει ταξινομηθεί θεωρείται έγγραφο που μπορεί να διαδοθεί από όποιον, να χορηγηθεί σε όποιον το ζητήσει. Δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί σε τράπεζες δεδομένων επίσης θεωρούνται τέτοιου είδους έγγραφα. Μπορούν, μπορεί να τα βρει κανείς από ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης. Αυτό ισχύει γενικότερα για τις δημόσιες διοικήσεις διεθνώς. Παράδειγμα, παίρνετε σημειώσεις μόνο σας από μία συνεδρίαση, αυτό δεν είναι έγγραφο. Αν όμως γίνει έγκριση και ψηφιστεί από τους συναδέλφους σας, τότε γίνονται οι σημειώσεις αυτές έγγραφο. Ο ορισμός αυτός είναι πολύ ευρύτερος από τον περιορισμένο των επισήμων εγγράφων όπως χρησιμοποιείται στα κράτη-μέλη και είναι πολύ κοντύτερα στην έννοια που δίνει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία στον όρο πληροφορία. Έχω ακούσει πολλά επιχειρήματα για το καλύτερο ορισμό και αν συμφωνούμε ότι χρειάζεται σαφέστερος από τον ισχύοντα νομίζω ότι ο καινούριος που δίνουμε είναι ικανοποιητικό. Δεύτερον, η εξισορρόπηση μεταξύ δικαιώματος πρόσβασης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να συνδυάσουμε τους κανόνες με τη, για τη δημόσια πρόσβαση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που προτείνει ο κανονισμός 45 του 2001. Δεν είναι δυνατόν το 1049 να το αποσυνδέσουμε τελείως από το 45. Προτείνουμε λοιπόν μία σε δύο βήματα να γίνει η διόρθωση πρώτον τα ονόματα και οι θέσεις των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και οι δραστηριότητές τους πάντοτε μπορούν να δοθούν σε όποιον τα ζητήσει. Ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι 90 με 95% των περιπτώσεων αίτησης πληροφόρησης αυτό αφορούν. Αν υπήρχε αυτή η πληροφόρηση δεν θα είχε υπάρξει υπόθεση Λάγκερ στο δικαστήριο. Δεύτερη φάση θα απαιτείται παρόλα αυτά έλεγχος για το κατά να απειλείται ή ο ιδιωτικός χαρακτήρας της πληροφόρησης που ζητιέται. Και τρίτον, η πρόσβαση στα έγγραφα που προέρχονται από τις χώρες μέλη. Η πρόταση της Κομισιόν απλώς κωδικοποιεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στη λεγόμενη υπόθεση INFOP από το 2005, το Δεκέμβριο του 2005. Γιατί ορισμένε φορές θεωρείται ότι υπάρχει δικαίωμα βέτο από τα κράτη-μέλη για τη χορήγηση πληροφόρηση, αλλά το δικαστήριο αυτό το απαγόρευσε. Πολλές φορές τα κράτη-μέλη απλώς αρνούνται να χορηγήσουν πληροφόρηση. Τώρα θέλαμε να κωδικοποιήσουμε νομικά το εξής. Εάν ένα κράτος μέλος δεν θέλει να χορηγήσουμε ένα από τα έγγραφα που μας έχει υποβάλει θα πρέπει να, το δικαιολογεί, να δικαιολογεί την άρνησή του. Και η δικαιολογία θα πρέπει να συμφωνεί με τον κανονισμό 1049. Τέλος, οι προσωρινές απαγορεύσεις στην πρόσβαση σε πληροφόρηση κατά τη διάρκεια ερευνών η πρόταση της Κομισιόν αποσαφηνίζει ότι απαγορεύεται η χορήγηση η πληροφόρηση όσο διαρκεί κάποια έρευνα. Γιατί είναι προφανές ότι στη διάρκεια, κατά τη διάρκεια μιας έρευνας μπορεί η χορήγηση των πληροσχετικών πληροφοριών να βλάψει ένα από τα δύο ή περισσότερα μέρη. Αλλά η πρόσβαση μπορεί να δοθεί όταν λήξει η έρευνα και αφού εφαρμοστούν ή σχετικές αποφάσεις. Ήδη συμβαίνει αυτό σήμερα. Αλλά επειδή δεν έχει κωδικοποιηθεί χρειάζεται πολύ περισσότερη γραφειοκρατία και κοστίζει περισσότερο και στον χρήστη. Το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν θα είναι το ίδιο αλλά θα είναι πιο σαφές νομικά και ελαφρύτερο γραφειοκρατικά. Και ερωτώ τώρα, σε πόσες χώρες μέλη επιτρέπεται η χορήγηση πληροφόρηση κατά τη διάρκεια μιας έρευνας σε καμία. Και για να αποδείξουμε ότι δεν παραμένουμε στα λόγια, αναφέρω ότι τον περασμένο Ιούνιο την επίσημη μου αλληλογραφία την υπέβαλα στην ιστοσελίδα μου. Είναι διαθέσιμη. Καλύτερα μητρώα, μεγαλύτερη φιλικότητα προς τον χρήστη και προσβασιμότητα και συντομότερη δημοσίευση των επισήμων εγγράφων. Υπάρχει ας πούμε η ιστοσελίδα που δίνουμε στους λομπιίστες που δείχνει πόσο αποτελεσματικά είναι όλα αυτά γιατί αποτελούν τμήμα της ευρωπαϊκής ιδέας για τη διαφάνεια. Αυτή είναι η κυρίαρχη αρχή. Το δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει διαφάνεια πρόσβαση. Νομίζω ότι τις ίδιες ιδέες θα τις έχετε ακούσει και στα κράτη-μέλη. Αυτό αναμένουν οι πολίτες εξάλλου. Τώρα έχω αναλάβει την πρωτοβουλία να σας απαριθμίσω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εκτός από αυτά τα τέσσερα που σας ανέφερα. Τους επόμενους μήνες θα συζητήσουμε με τα άλλα θεσμικά όργανα ένα σχέδιο δράσης για την ανοιχτή πρόσβαση, γιατί πρέπει να πάρουμε μαθήματα από πρακτικά παραδείγματα. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Και τώρα ανοίγει η συζήτηση. Έχω επτά ονόματα στο κατάλογο. Συνήθως έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας. Τέσσερα το πολύ. Εντάξει, είναι τόσο ανεκτών ορίων αυτό. Πρώτος ο Τζάκομο Σαντίνη από την Ιταλική Γερουσία και ακολουθεί ο Μπόγκταν Τζέμιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, προσωπώ την Ιταλική Γερουσία. Με μεγάλη προσοχή άκουσα τις βασικές παρατηρήσεις στον παλιό μου συνάδελφο τον κύριο Κάσμαν και την κυρία Επίτροπο. Άκουσα τις νέες ιδέες που προέκυψαν μετά από όλα αυτά τα χρόνια των συζητήσεων που καμιά φορά ήταν και δημαγωγικές συζητήσεις. Το άρθρο 42 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είναι σαφέστατο. Βέβαια, από την άλλη, η καθημερινή του εφαρμογή, ο περίφημος ε, διαθεσμικός διάλογος υπολείπεται κατά πολύ. Η Επίτροπος ε, υπέβαλε ορισμένε ε, ερωτήσεις και εγώ έχω να ερωτηθεί πολλές φορές. Σε τι χρησιμεύει η διαφάνεια την οποία επικαλούμαστε. Ποιοι είναι οι πολίτες που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα και ποιος είναι ο στόχος μας. Πρώτος στόχος βεβαίως η διοικητική διαφάνεια, προφανής. Τι σημαίνει αυτό όμως συγκεκριμένα. Είναι μια υπηρεσία που προσφέρουμε στους πολίτες και στους εκπροσώπους τους. Άρα και στους βουλευτές και στα ίδια τα θεσμικά όργανα. Είναι μια υπηρεσία, είμαστε στην υπηρεσία των πολιτών και ε, τα θεσμικά όργανα έχουν συμφέρον να γνωρίζουν γι' αυτά οι πολίτες και να τους εκτιμούν. Από την άλλη όμως υπάρχει ορισμός του πολίτη. Ποιος είναι πολίτης. Υπάρχουν μια σειρά φορέων εδώ, αλλά και θεσμικά όργανα που έχουν θεσμικό διάλογο μεταξύ τους. Και πού είναι αυτή η συνοχή, προς το παρόν όνειρο και μόνο είναι. Όταν όμως εφαρμόζονται όλα αυτά σωστά, ε, μας εμπιστεύεται ο πολίτης και συμμετέχει στην προσπάθειά μας και συμμερίζεται και τα ιδανικά μας για να έχουμε τελικά ε, εμπλουτισμένη δράση στην υπηρεσία πάντα των πολιτών. Και νομίζω ότι ότι μάλλον δεν θα πρέπει να συμβεί στους νέους βουλευτές. Θεωρώ ότι ο βουλευτής ορίζεται από τους, από τους ε, ψηφοφόρους του για να διεκπαιρεώσει ένα συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, φέρει συγκεκριμένη ευθύνη έναντι των πολιτών και θα πρέπει να βρίσκεται άνω των άλλων θεσμών ή θεσμικών οργάνων. Και πολλές φορές αυτό που θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει μια στρεβλωμένη χρήση ευαίσθητων εγγράφων, αυτό είναι θεμικό, θεμητό. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που μπορείτε να αρνηθείτε στο μεμονωμένο πολίτη δεν μπορείτε να το αρνηθείτε στον βουλευτή. Ο βουλευτής θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, ακόμα και εμπιστευτικού χαρακτήρα, γιατί είναι σίγουρο ότι ο βουλευτής μπορεί να διαχειριστεί το ζήτημα πολύ καλύτερα, με την, ε, με την διακριτική του ευχέρεια, με διάβια και ούτω καθεξής. Εγώ βρίσκομαι εδώ για ε, δύο θητείες. Πολλές φορές ε, για να ζητήσουμε απλές πληροφορίες για ένα φάκελο πρέπει να περάσουμε από 40 κύματα. Ερχόμαστε σε επαφή με έναν απλό υπάλληλο της Κομισιόν και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να ζητήσω από την FBI την προσωπική διεύθυνση του Μπιν Λάντεν από το να ζητήσω μια πληροφορία από έναν υπάλληλο της Κομισιόν. Άκουσα λοιπόν από την Επίτροπο και αυτά είναι δικά της ε, λόγια, ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην Επιτροπή. Ελπίζω ε, αυτό να μην ε, παραμείνει επί χάρτου, αλλά να αποτελέσει καθημερινότητα στις σχέσεις μας με τα άλλα θεσμικά όργανα. Και αυτό ιδιαίτερα για τους βουλευτές, αλλά θα πρέπει να ισχύει για όλα τα επίπεδα. Δηλαδή από τον Επίτροπο μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο δηλαδή η προσπελασιμότητα, η πρόσβαση στα έγγραφα. Διότι δεν γίνεται για λόγους νοσηρής περιέργειας, αλλά αντικατοπτρίζει την ευθύνη του έναντι των πολιτών. Και όταν ο πολίτης δεν έχει επαρκείς πληροφορίες και δεν έχει και τη δυνατότητα προσβασιμότητας, τότε θα πρέπει να παρέμβει ο βουλευτής θα πρέπει να παρέμβει για να εξασφαλίσει αυτές τις ε, πληροφορίες. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε νέες κατευθυντήριες γραμμές για να φτάσουμε όχι μόνο στην διάβγεια αλλά και στην αποτελεσματικότητα των σχέσεών μας. Θα πρέπει να συντονίσουμε τη μέθοδο πρόσβαση στα έγγραφα με κοινέ κατευθυντήριες γραμμές. Μας είπε ο κύριος ε, Κάσμαν ε, με μεγάλη διάβγεια και ανάλογα με τον τύπο του εγγράφου. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κοινέ κατευθυντήριε γραμμές για τι σχέσει των θεσμικών οργάνων. Δηλαδή, όταν μιλάμε για προσπελασιμότητα μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής θα πρέπει να είναι του ίδιου χαρακτήρα όπως ισχύει και στις εθνικές διοικήσεις στους Δήμους και στις περιφέρειες. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε task force που να μπορούν να οργανώσουν αυτή την κοινή εργασία. Να μιλάμε την ίδια γλώσσα και να μπορέσουμε να επιταχύνουμε και τους ε, χρόνους. Πρόκειται για προτάσεις που ίσως φαίνονται ουτοπικές, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που κατέδειξαν ότι υπάρχει κοντοθορισμός πολλές φορές στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Υπάρχει δυσπιστία, άσκοπη δυσπιστία και νομίζω ότι αυτό θα ήταν ο τελευταίος στόχος τον οποίο θα επιθυμούσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαντίνη. Uh, Η κυρία Ριπέλοβα έχει το λόγο και τώρα έχει το λόγο ο κύριος ε, ένας βουλευτής από την Σλοβενία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζουμε τις προθέσεις ε, της ε, Επιτροπής να αλλάξει την οδηγία, λέει ο κύριος Τσέπιτς, και θα θέλαμε να είμαστε σίγουροι ε, ως προς τις ε, επιπτώσεις της οδηγίας και να υπάρχουν ε, και να υπάρχει μια ευρύτερη προσπελασιμότητα ως προς την εμβέλεια αυτή και την πρόσβαση χωρίς να μειώσουμε τον κανονισμό. Δηλαδή, καλωσορίζουμε τις προθέσεις της Επιτροπής ε, που αναφέρει ότι θα πρέπει να ορίζουμε όλες τις εξαιρέσεις σε μία και μεμονωμένη πράξη. Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην εφαρμογή του κανονισμού 1049, διότι η μεταφορά αυτή στο, στην εθνική ένομη τάξη δεν θα πρέπει να αλλάξει την εμβέλεια των, και των δύο κανονισμών. Βεβαίως, ο κανονισμός του άρχους και ο κανονισμός 1049 έχουν ε, διαφορετικό σκεπτικό και εμβέλεια. Η Σλοβενία έχει μία συγκεκριμένη θέση που συνάδει με τη θέση άλλων κρατών μελών. Η Σλοβενία επίσης έχει την ε, ίδια άποψη με τα κράτη τα οποία τονίζουν την ειδική χρήση αυτών των ορισμών. Θα θέλαμε να συλλέξουμε όλες τις εξαιρέσεις σε ένα άρθρο και την δυνατότητα να μπορέσουμε να ορίσουμε νέα κατηγορία εγγράφων που θα είναι δημόσια έγγραφα. Επίσης θα θέλαμε να μεγαλώσουμε την εμβέλεια και την ε, προσβασιμότητα σε αυτά τα έγγραφα. Υπάρχουν ορισμένα ασαφή ζητήματα σε σχέση με τις αποφάσεις. Για παράδειγμα, όταν το θεσμικό όργανο έχει ε, ορισμένες ε, εξηγήσει, αλλά δεν τις θεωρεί επαρκείς. Σε αυτήν την περίπτωση ο ετών έχει τη δυνατότητα να ζητήσει κάποιο είδος ανταπόδοσης για αυτή την άρνηση. Η Σλοβενία θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα γενικά, αλλά η πρώτη παράγραφος του άρθρου 12 θα πρέπει να παραμείνει ως έχει, διότι ενέχει και το, την αιτιολογική σκέψη των θεσμικών οργάνων για να υπάρχει ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα έγγραφα. Όμως, ο στόχος της διεύρυνσης αυτής μπορεί να οδηγήσει σε άλλο διοικητικό φόρτο για τα θεσμικά όργανα. Θα πρέπει επίσης να προστατεύουμε τα νομικά πρόσωπα, διότι το θέμα της ασφάλειας δικαίου σχετίζεται πολλές φορές και με φυσικά πρόσωπα. Επίσης, καλωσορίζουμε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συλλέξει όλους τους κανόνες σε μία ενιαία πράξη αλλά συμμεριζόμαστε και την άποψη των χωρών που θεωρούν ότι η εξαίρεση δεν είναι σαφής και θα πρέπει να το επανορθώσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ριπέλοβα από την Τσεχία και μετά ο Λόρτ Bones. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή την συζήτηση και θα ήθελα να σας πω ποια είναι η θέση της τσεχικής γερουσίας σε σχέση με την ε, αναθεώρηση του κανονισμού για την πρόσβαση σε έγγραφα. Το συζητήσαμε στις 3 Οκτωβρίου στη Γερουσία και φτάσαμε σε μία απόφαση όπου καλωσορίζουμε την ε, προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της προσβασιμότητας αυτής, αλλά η τσεχική γερουσία θεωρεί ότι αυτή η πρόταση αποτελεί οπισθοδρόμηση ως προσορισμένες αρχές, γιατί δεν προβάλλει την νομιμότητα καθώς και τη λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το κοινό. Θεωρούμε ότι ο ορισμός, οι ορισμοί υπάρχουν, αλλά δεν είναι αρκετά ευρύς, έτσι ώστε να υπάρχει σωστή πρόσβαση στα έγγραφα, διότι η πρόσβαση θα ήταν χειρότερη αν λάβουμε υπόψη αυτό τον ορισμό. Και η Γερουσία λυπάται ιδιαίτερα διότι η πρόταση δεν αυξάνει την ε, διαφάνεια των μητρών των διαφόρων θεσμικών οργάνων και την ε, διασυνδεσιμότητά τους. Όπως ξέρετε, υπήρξε μια αντίδραση και στις 6 Ιανουαρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υπερασπίζεται τον ορισμό της και θεωρεί ότι η πρόθεση δεν ήταν να μειωθεί ο όγκος των εγγράφων ή ο τύπος των εγγράφων, αλλά ορίζει το ότι το έγγραφο θεωρείται έγγραφο όταν λάβει τελική μορφή και αποσταλεί σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς δικαιούχους. Θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας για μια κοινή πύλη ως προς την πρόσβαση στα κοινά αυτά μητρώα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπη για τις επαυτές αυτές με τα Εθνικά Κοινοβούλια και θεωρώ ότι η πρόταση αυτή θα εγκριθεί κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη του κοινού. Ωραία, τώρα θα συνεχίσουμε με τον ε, Lord Bones και μετά ε, με τον κύριο Μαουρίτσιο Τούρκο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και την Επιτροπή και την Τσεχική Προεδρία που οργάνωσε αυτή τη συνεδρίαση που έχει μεγάλη σημασία μέσα στα πλαίσια και της δικής μας υποεπίτροπης που ασχολείται με αυτό το ζήτημα, διότι εξετάζουμε αυτή την ε, προτινόμενη, αυτή την πρόταση κανονισμού. Η διάβγεια είναι αναπόσπαστο θέμα και ζωτική σημασίας για την πίστη των, ε, του κοινού και για τη λογοδοσία μας. Και νομίζω ότι όλα τα κοινοβούλια θα εγκρίνουν την έκθεση Κάσμαν για να υπάρχει ε, μεγαλύτερη και καλύτερη προσπελασιμότητα. Μιλάμε λοιπόν για διάβια και χωρίς να προσκρούσουμε στη, σε θέματα ε, ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτικού βίου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι Εάν δεν μπορούσε το κοινό να έχει αυτή την πρόσβαση, αυτό θα ήταν ε, ιδιαίτερα ε, βλαβερό και ζημιογόνο και θα φτάναμε σε, ένα, σε μια σκοταδιστική, ε, σκοταδιστικό ορισμό του ζητήματος σε σχέση με τις συμβουλές που παρέχονται. Θα ήθελα να τονίσω το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και το εποπτικό τους καθεστώς με βάση την πείρα μου στη δική μου επιτροπή. Πρόσφατα εγκρίναμε μία πρόταση για την κοινοτική νομοθεσία και θεωρούμε ότι η διαδικασία είναι αρκετά ανοιχτή για αυτούς που θέλουν να, ακολουθήσουν, να παρακολουθήσουν αυτές τις εργασίες. Το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής δεν αποτελεί καθαρή εξουσία. Αυτό είναι μύθος διότι μπορεί να προτείνει αλλά δεν μπορεί να αποφανθεί κάτι το οποίο μπορεί να κάνει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, έρευνας Είδαμε και το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων ως προς τη λογοδοσία των κυβερνήσεών τους και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να είναι πιο δραστήρια στη διαμόρφωση της νομοθεσίας και ως προς την ανταπόκρισή μας στα έγγραφα της Επιτροπής. Η πρωτοβουλία του Πρόεδρου Μπαρόζο ήταν πολύ καλή, δηλαδή το ότι αποτάνθηκε απευθείας στα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτά τα θέσαμε σε εφαρμογή με βάση την πράσινη βίβλο της Επιτροπής. Δώσαμε μία απάντηση και ζητήσαμε έναν ενιαίο κώδικα έτσι ώστε να προωθήσουμε την διάδοση των πληροφοριών. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένοι περιορισμοί, ιδιαίτερα για σημαίνοντα ζητήματα, αλλά το δικαίωμα των ατόμων θα πρέπει να προωθηθεί με βάση τον παρόντα κανονισμό ιδιαίτερα ως προς τον εμπιστευτικό χαρακτήρα για εμπορικά ζητήματα. Θεωρώ ότι τα εθνικά κοινοβούλια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως προς τον έλεγχο, εποπτεία και λογοδοσία. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μία εξισορρόπηση μεταξύ διαφάνειας και άλλων νομικών ή νομοθετικών διαδικασιών. Ίσως, ίσως είναι δύσκολο να γίνει αυτή η εξισορρόπηση, διότι εξαρτάται από τα συμφραζόμενα. Πολλές φορές οι κυβερνήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν θέματα ε, δικαστικών προσφυγών και θεωρούμε ότι μία ομάδα, μάλλον τα έγγραφα ομάδων εργασίας του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι δημόσια έγγραφα του Συμβουλίου. θα πρέπει να γίνει και μία διάκριση μεταξύ του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων για λόγους εποπτείας και μία προσέγγιση πέρα από τα σύνορα. Και αυτό αφορά και την αποκάλυψη εγγράφων, τη διάδοσή τους μετά από την έγκρισή τους. Και θα πρέπει να γίνει μία διάκριση μεταξύ ε, των ε, συμβουλών και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ε, αντιμαχόμενα μέρη. Αυτή νομίζω ότι θα ήταν και μία ε, ισορροπημένη προσέγγιση. Ευχαριστούμε τον Λόρδο Bones και το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μαουρίτσιο Τούρκο. Και μετά ο κύριος Αρκάδιο Ντίας Τεχέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον ε, πρόεδρο Ζεράρ Ντεπρέ της Επιτροπής ε, Πολιτικών Ελευθεριών και το Κοινοβούλιο της Τσεχίας που διοργάνωσαν αυτές τις συνεδριάσεις. Βεβαίως, τα σχόλια του κυρίου Κάσμαν, καθώς και η παρέμβαση της κυρίας Βάλστρομ, είναι ε, άκρος σημαντικές σε σχέση και με τις πρόσφατες εξελίξεις διότι όλα αυτά δεν είναι κεκτημένα, δεν είναι δεδομένα για τους πολίτες αλλά και για τους βουλευτές, τους εθνικούς βουλευτές. Ο συνάδελφος από το Ηνωμένο Βασίλειο θεώρησε ως δεδομένο ότι στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης είναι διαθέσιμα στους ε, βουλευτές. Αυτό δεν ισχύει ή μάλλον δεν ίσχυε μέχρι λίγους μήνες πριν. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω το Βασίλειο της Σουηδίας που δέχτηκε τη δική μου προσφυγή ενώπιον του ΔΕΚ ζητώντας δημοσιότητα της, των ε, καθαρά νομικών συμβουλών, συμβουλών νομικού χαρακτήρα. Και το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βασίλειο της Σουηδίας και η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου ε, ζήτησαν κάτι παρόμοιο γιατί δεν ήθελαν να κοινοποιούνται οι νομικές γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά την απόφαση του ΔΕΚ, όπου 13 ε, δικαστές ομόφωνα ε, απέρριψαν αυτά τα δεδομένα και είπαν ότι πρέπει να αλλάξει η τάξη πραγμάτων, ο σύγχρονος Νομπράουερ εκπροσώπησε πάρα πολύ καλά τον έναν διάδικο, δηλαδή εμάς. Και τώρα, με την αναθεώρηση του κανονισμού για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη ερμηνείας, τα οποία μας ε, δίπουν όλα αυτά τα χρόνια. και τα οποία ακύρωναν τα θετικά αποτελέσματα ή τις καινοτομίες που πρότειναν οι κανονισμοί. Αυτό που σήμερα ο κύριος Σολάνα θεωρεί απόρριτο ή άκρος απόρριτο και κλεισμένων των θυρών, ίσως να μην έχει και μεγάλη σημασία ή να έχει σημασία, ε, γιατί ένας από τους 27 ε, υπουργούς εξωτερικών το διαψεύδει. Αλλά ό,τι περνάει και από το γραφείο του κυρίου Σολάνα δημοσιοποιείται εν ευθέτω χρόνο και διατίθεται στους βουλευτές. Σε θεσμικό επίπεδο όμως δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος, πλήρης δημοκρατικός έλεγχος, γιατί σε κάθε κράτος υπάρχει μια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία μπορεί να προωθήσει έρευνες και σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μπορεί να ζητήσει με ευγένεια ορισμένα έγγραφα και αν ε, τα αρνηθούν τότε ίσως θα πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη από πάνω. Σε σχέση με τον νέο κανονισμό και τον συνάδελφο Κάσμαν που ήταν ε, ο φρουρός του Κοινοβουλίου, η εμπροστοφυλακή μπορώ να πω για την προσβασιμότητα στα έγγραφα, ε, ορίζει ότι στα πλαίσια του ορισμού θα πρέπει να υπάρχει και η έννοια της ε, πληροφορίας, όπως γίνεται και στη ΣΥΠΑ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενσωματώσουμε μία ρήτρα όπου σε περίπτωση παράληψης των θεσμικών οργάνων θα πρέπει ε, να γίνεται άμεση ε, δημοσιοποίηση. Ο κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει όλα τα έγγραφα, όχι αυτά ε, που έχουν νομικό χαρακτήρα ή νομοθετικό χαρακτήρα. Και μέσα στα πλαίσια της επιτροπολογίας και στα πλαίσια της πρώτης ανάγνωσης και του τριμερούς διαλόγου. Θα πρέπει να έχουμε ανοιχτή πρόσβαση και να υπάρχει ένα καθεστώς πολυγλωσσίας με έναν ελάχιστο παρονομαστή όπως ορίζουν οι συνθήκες. Αυτό ισχύει και για τα μητρώα, για τα μητρώα μας. Στην προηγούμενη θητεία οι δραστηριότητες του Προέδρου της Επιτροπής καθώς και η ελογραφία του ε, βρισκόταν στο διαδίκτυο. Σήμερα δεν υπάρχουν πια αυτά τα δεδομένα. Θα πρέπει επίσης να περιορίσουμε τις εξαιρέσεις όπως ο εμπιστευτικός χαρακτήρας νομικών γνωμοδοτήσεων και επίσης να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα τα κράτη-μέλη ως προς τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να σας σταματήσω γιατί έχετε υπερβεί το χρόνο σας. Σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια και τη θέση τους ε, στο Συμβούλιο Υπουργών θα μιλήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε το εξής. Κατά πόσο για να γνωρίζουμε τη θέση των εθνικών αντιπροσωπιών θα πρέπει να αποτανθούμε στο ΔΕΚ ή μπορεί αυτό το ζήτημα να έχει μια πολιτική λύση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τούρκο και τώρα Δίνω τον λόγο στον κύριο Αρκάτιο Ντίας Τεχέρα από την Ισπανική Γερουσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Οι κρατικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ισότητα ε, και την ισονομία όλων των πολιτών και να ε, προωθούν τη συμμετοχή όλων στην πολιτική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή. Αυτό είναι ένα άρθρο του Ισπανικού Συντάγματος από το έτος 1978 και ε, υπάρχει το γερμανικό και το ιταλικό που αντίστοιχα ε, μιλούν γι' αυτό. Μπορεί να είναι ουτοπία, αλλά είναι στόχος πραγματικά στην ουσία ε, να λέμε αυτό που μας ενδιαφέρει να υπάρχει μόνιμη δουλειά με επιμονή να είμαστε προσυλλομένοι σε αυτό το στόχο της ισότητας όλων των ανθρωπίνων όντων και το καθεστώς του πολίτη. Άνδρας και γυναίκα πολίτης έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη γνώση. Εδώ πριτανεύει ο όρος αξιολόγηση. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Κάσμαν, την κυρία Βάλστον και βλέπω ότι υποβόσκει εκεί ένα πάθος κάτω από τις παρεμβάσεις αυτές για το στόχο αυτό ε, που μας ε, εμπνέει όλους να είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στην πρόσβαση στη γνώση. Επτά χρόνια λοιπόν και αξιολόγηση της πορείας και μου έκανε εντύπωση κυρίως ότι ε, τα πανεπιστήμια και οι ομάδες πίεσης ενδιαφέρονται περισσότερο για τα θέματα αυτά. Και ρωτώ, ποιο είναι το ποσοστό των πολιτών που ενδιαφέρεται βέβαια με σχετικούς όρους στην πρακτική καθημερινή δουλειά, διότι καμιά φορά κύριε Κάσμαν έχω την εντύπωση ότι ο Δον Κιχώτης είναι ε, στη, στους νόμους, ενώ στην καθημερινή ζωή είναι ο Σάντσο Πάντσα. Και εγώ, όπως βλέπετε, μοιάζω έτσι σωματικά με το Σάντσο Πάντσα. Μπορεί να έχω στο μυαλό μου το Δον Κιχώτη, αλλά στην καθημερινή ζωή ως Σάντσο Πάντσα θα πρέπει να βλέπω πώς εφαρμόζονται οι νόμοι. Γιατί νόμοι χωρίς εποπτεία, χωρίς παρακολούθηση, χωρίς δράση τελικά είναι ευσεβής πόθη, ρητορική, κενό γράμμα και φιλολογία ωραία ή λιγότερο ωραία αλλά δεν είναι η ενσάρκωση των δικαιωμάτων στην καθημερινότητα του πολίτη. Λοιπόν, διαρωτούμε, μήπως σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, την προληπτική και τις δράσεις, ε, να προχωρήσουμε σε μια εκπαίδευση των πολιτών που λέμε χτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ε, είναι εκπαίδευση των πολιτών. Γιατί? Υπάρχει αυτό το καθεστώς του Ευρωπαίου πολίτη, του πολίτη που είναι όλοι ισότιμοι μεταξύ τους και ελεύθεροι. Αλλά αν δεν έχουν δικαίωμα στη γνώση και δεν έχουν οδούς να φτάσουν μέχρι τη διαφάνεια, όλα αυτά που τους λέμε είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά ρητορίες. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πραγματικά ένα σχολείο διαπαιδαγώγησης, αγωγής του πολίτη, ε, καθημερινά, ναι. από όλα τα θεσμικά όργανα. Όλοι μιλάμε εδώ για προδιαγραφές, για απαιτήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να είναι καθημερινή μας πράξη στι χώρες μα. Αυτό μου φαίνεται σημαντικό εμένα. Ε, ζήτημα δεύτερο τώρα. Υπάρχει εμπειρία κοινοβουλευτική, όπου πραγματικά οι βουλευτές έχουν πρόσβαση ε, στην ενημέρωση, ε, πρόσβαση που δεν έχουν οι πολίτες και η συνάδελφος ε, που είναι δικηγόρος από την Ισπανική Βουλή υπάρχει μια ε, επιτροπή ε, απορρίτων όπου συμμετέχουν οι γραμματείς των πολιτικών ομάδων, των κομμάτων και έχουν πρόσβαση εκεί βουλευτές, πρόσβαση στην οποία δεν μπορούν να καταφύγουν πολίτες. Ας πούμε, στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Έχουμε πληροφοριοδότες που δεν ε, θέλουν το όνομά τους να δημοσιοποιείται, ούτε καν προς τους βουλευτές, ούτε έχουν συμφέρον γι' αυτό. Άρα, λοιπόν, υπάρχει μια διαβάθμιση και μια εμπιστευτικότητα σε αυτές τις πληροφορίες, αλλά οι βουλευτές τις βλέπουν. Στη συνέχεια, τρίτο, Υπάρχει μια σύγκρουση εδώ δικαιωμάτων. Μιλάμε για ένα θεμελιώδες δικαίωμα που είναι το δικαίωμα στην πρόσβαση, αλλά υπάρχει και άλλο θεμελιώδες δικαίωμα που είναι η προστασία των δεδομένων. βιομηχανική ε, ιδιοκτησία, ανήλικη, ασφάλεια, άμυνα. Όταν συγκρούνται λοιπόν δύο δικαιώματα τέτοια θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το πιο αξιοσέβαση, ποιο αξίζει περισσότερο μάλλον προστασίας. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα γενικό κανόνα απόλυτο. Όταν ε, θες να έχεις πρόσβαση να έχεις. Ε, θα πρέπει κάθε φορά να σταθμίζουμε με βάση την προηγούμενη ε, πρακτική και όχι τη ε, ρητορία και τις διακήρυξεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την επίοικιά σας και την καλοσύνη σας. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας το Δον Κιχώτη πάντα, αλλά καθημερινά να έχουμε την παρακολούθηση και το μάτι του Σάντσο Πάντσα. Αλλιώς οι προδιαγραφές είναι διαφορετικές στην Ευρώπη ας πούμε ε, και στις χώρες μας. Αυτό που απαιτούμε από την Ευρώπη και αυτό που απαιτούμε από τις χώρες. Θα πρέπει τα θεμελιώδη δικαιώματα και η καθημερινή μας νομική πράξη να συνάδει. Όπου και αν είμαστε Ευρωπαίοι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Επόμενος ομιλητής, ομιλήτρια, η κυρία Γκραμπόφσκα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Τσεχική Προεδρία και την ε, Επιτροπή υπό την αιγίδα του κυρίου Ντεπρέ που μας έδωσε την ε, δυνατότητα να συνεδριάσουμε για αυτά τα θέματα ύψης της σημασίας. Όλοι ξέρουν γιατί ακριβώς μιλάμε, διότι επανερχόμαστε σε αυτά τα θέματα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων. Αυτό το θέμα μας έχει απασχολήσει ε, μακρόν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υπάρχει μία εξισορρόπηση στα έγγραφα αυτά και στην πρόσβαση στην πληροφορία υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια. Πέρα δηλαδή από την ε, πρόσβαση στα έγγραφα αυτά, στρίκτο σένσου. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ανισορροπία μεταξύ αυτών των ε, δύο ενιών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρόσβαση στα έγγραφα αυτά για τους εθνικούς βουλευτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διευρυνθεί ως έννοια τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της Λισαβόνας και τη στιγμή που μιλάμε για την αντίδραση των ε, εθνικών κοινοβουλίων σε σχέση με τα έγγραφα που προετοιμάζει το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι η συνθήκη της Λισαβόνας μας ε, επιτρέπει την πρόσβαση στα έγγραφα και δεν μιλάμε για αποκλειστικό δικαίωμα των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά και υποχρέωση αντίδρασης των εθνικών κοινοβουλίων στα πιο σημαντικά ζητήματα που θίγουν αυτά τα έγγραφα. Ε, αντίδραση και προς τα τρία θεσμικά όργανα. Θα ήθελα να τονίσω και μία άλλη πτυχή του ζητήματος τις ευθύνες μας έναντι των συμπολιτών μας. Συνέταξα μία έκθεση για το ρόλο της κοινωνίας μέσα στα πλαίσια του διαλόγου με τον πολίτη. Και υπάρχει ένα ζήτημα κλειδί. Ζήτημα κλειδί που αφορά την επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτη. Αυτό θα, σε αυτό θα υποβοηθήσουν και τα εθνικά κοινοβούλια και όχι μόνο το ευρωπαϊκό, ε, έτσι ώστε να διαδίδονται οι πληροφορίες και να φτάνουν στο τελικό αποδέκτη όχι μόνο με μεσολαβητή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εδώ ο, ο ρόλος μας είναι πολύ μεγάλος θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις πλέον πρόσφατες τεχνικές πολυμέσων έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να έχουν εύκολη πρόσβαση ε, μέσω διαδικτυακών πυλών. Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσε να μας προσάψει κανείς τίποτα, ότι δηλαδή παρακολύουμε την διάδοση των πληροφοριών. Θα ήθελα οι επόμενοι ομιλητές να τηρήσουν τα τρία λεπτά, αυστηρά τα τρία λεπτά. Η κυρία Μωρέ Σαρμέντο από την Πορτογαλική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κύριε Σαρμέντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα συμμετοχής σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήματα που σχετίζονται με το δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα. Η αιτιολογική σκέψη 16 αναφέρει ρητός ότι ο παρόν κανονισμός δεν προδικάζει την προσπελασιμότητα σε εθνικά έγγραφα και μέσα στα πλαίσια μιας δικαστικής έρευνας. Και οι δύο βασικοί δικαιούχοι γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι, αλλά ο τελικός ε, δικαιούχος είναι οι πολίτες. και αυτό αφορά όλα τα κράτη-μέλη, τους πολίτες όλων των κρατών μελών. Το ερώτημά μου έχει ήδη τεθεί, αλλά εγώ θα ήθελα να μιλήσω και για μία άλλη κατηγορία, μία άλλη κατηγορία πολιτών που είναι οι δημοσιογράφοι. Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα αφορά όλες τις χώρες και είναι γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι ανεξάρτητα από το λειτουργήμα και τις υποχρεώσεις του, υποχρεώσεις τους που πρέπει να πληροφορούν το κοινό, ζητούν ε, συνεχή ροή πληροφοριών και ζητούν ε, άλλα προνόμια, πέρα δηλαδή από αυτά που έχει ο απλός πολίτης. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο και αυτοί ε, συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των ε, δικαιούχων. Σε σχέση με τα έγγραφα κάθε αυτά, όπως ξέρετε η Πορτογαλία έχει μεταφέρει την οδηγία, δηλαδή την προγενέστερη οδηγία του 2003 και αναφέρεται ε, ρητά στην νέα πρόσβαση στα έγγραφα ως προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί κανείς μετά την ε, αίτηση να υποβάλει και μία αιτιολόγηση ή μπορούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να χρησιμοποιήσουν αυτά τα έγγραφα για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που έχουν αναφερθεί αρχικά. Ε. Σας ευχαριστούμε για την ερώτηση και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Μόργαν Γιώχανσον από τη Σουηδία και μετά ο Μάρκο Καπάτο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Είμαι ο Μόργαν Γιώχανσον, συμμετέχω, είμαι βουλευτή στη Βουλή των Αντιπροσώπων Σουηδία. Ήμουνα γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ορισμένα χρόνια πριν και είχα ασχοληθεί με τον αρχικό κανονισμό δημόσιας πρόσβασης που αποφασίστηκε κατά τη Σουηδική Προεδρία το 2001. Και θεωρώ ότι οι αποφάσεις του 2001 δεν ήταν καινοτόμες σε σχέση με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα γίνεται μία ανακεφαλαίωση αυτών των ε, κανονισμών και έχουν προταθεί ορισμένες αλλαγές. Ε, γίνονται, λοιπόν, υπάρχουν αλλαγές ε, που πραγματικά βελτιώνουν το καθεστώς της διαφάνειας, όμως δυστυχώς υπάρχουν και θέματα που αποτελούν μία παλινοδία σε σχέση με την διαφάνεια. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ως προς τον ορισμό του δημοσίου εγγράφου ε, έχουμε μια πιο συσταλτική, έναν πιο συσταλτικό ορισμό. Έπειτα, ως προς ορισμένες κατηγορίες εγγράφων έχουν διευρυνθεί. Δηλαδή, λιγότερα εγγραφά θα ε, εμπίπτουν στο δικαιοδοτικό καθεστώς και πολλές φορές θα πρέπει να δούμε ότι προσκρούμε στην, ε, στην νομοθεσία που υπάρχει για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Άρα δεν υπάρχει πρόσβαση. Αυτό το έχει θίξει ο κύριος Διαμαντούρος, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο οποίος ε, είπε, ανέφερε ότι η πρόταση της Επιτροπής σημαίνει μικρότερη ε, πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άρα λιγότερη διαφάνεια και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μείζον μήνυμα. Υπάρχει συνένεση στη Σουηδία ότι ο κανονισμός αυτός έχει λειτουργήσει ε, πολύ καλά, αλλά αν γίνουν αλλαγές θα πρέπει να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια και όχι μικρότερη. Καλωσορίζω την παρουσίαση της κυρίας Βάλστρομ γιατί υπερασπίζεται την πρόταση αλλά δέχεται και τη δυνατότητα αλλαγών σε ορισμένα ζητήματα που ανέφερα. Αυτό ήταν ε, άκρος επικοδομητικό και ελπίζω κυρία Βάλστρομ να φτάσετε σε κοινή θέση με το Κοινοβούλιο επί αυτών των θεμάτων και αυτό θα ικανοποιήσει και τον ε, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ο κύριος Κάσμαν έχει συμμετάσχει σε αυτή τη ε, διαδικασία διαβουλεύσεων 10 χρόνια πριν. Ε, έχει πολύ επικοδομητική προσέγγιση και ελπίζω αυτά τα ζητήματα να διευθετηθούν κατά κάποιο τρόπο. Αυτό έχει σημασία και ευρύτερα. Η Ευρωπαϊκή, ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει να αντιμετωπίσει και ένα θέμα νομιμότητας καθαρά. Σε λίγους μήνες θα διενεργηθούν ευρωπαϊκές εκλογές και από όσο ξέρουμε Έγινε μια δημοσκόπηση στη Σουηδία και μόνο 40% των πολιτών θα συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές. Κάτι το οποίο αφορά και τα περισσότερα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να μειωθεί λοιπόν αυτό το χάσμα μεταξύ Ευρωπαίου πολίτη από τη μία πλευρά και ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό είναι ένα από του τρόπου για να το επιτύχουμε. Ευχαριστούμε ο κύριος ε, Μάρκο Καπάτο και μετά ο κύριος Σάση από το Φιλανδικό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Καπάτο, ευχαριστώ. Πρόεδρε, απλώς ήθελα να υπογραμμίσω κάτι που θεωρώ σημαντικό. Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα αποτελεί υπηρεσία, υπηρεσία προς τους πολίτες, όταν μιλάμε για μια νομοθετική διαδικασία καθαρά, δηλαδή μια διαργασία λήψης αποφάσεων, δεσμευτικών αποφάσεων, σε νομοθετικό πλαίσιο, εδώ περνάμε από την υπηρεσία σε μια υποχρέωση, απόλυτη υποχρέωση. Δηλαδή το θέμα της δημοσιότητας ε, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δημοκρατικής νομιμότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται και γι' αυτό νομίζω ότι οι πληροφορίες δεν είναι ε, τα έγγραφα, αλλά υπό την ευρύτερη έννοια οι πληροφορίες που αφορούν την νομοθετική διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν να μιλάμε για μια ε, δημόσια διαδικασία και η πρόταση επιτροπής αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιες είναι και οι συνέπειες της απόφασης ε, στην υπόθεση Τούρκο διότι το Συμβούλιο δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη αυτή την απόφαση σε σχέση με την ε, δημοσιοποίηση των αποφάσεων των ε, εθνικών αντιπροσωπιών. Με συγχωρείτε. Αυτά τα στοιχεία αποκρύπτονται από το Συμβούλιο. Γι' αυτό νομίζω ότι το Συμβούλιο στην πρότασή του που προετοιμάστηκε πριν από αυτή την απόφαση του ΔΕΚ ε, συρρυκνώνει την ερμηνεία της διαφάνειας, δηλαδή περιορίζεται στο άρθρο 255 της συνθήκης. Η Επίτροπος έχει δίκιο ότι μπορεί να γίνει τέτοια χρήση χωρίς να αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε μία έκθεση, δική μου έκθεση, όπου δεσμευόμαστε να καταγράφουμε ανοιχτά την παρουσία των Ευρωβουλευτών κατά τις ψηφοφορίες και στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια. Αλλά ο νόμος μπορεί να είναι χρήσιμος για να ξεπεράσουμε τα γραφειοκρατικά προσκόμματα. Και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να περιχαρακωθεί η διοίκηση πίσω από τεχνικές δίθεν δυσκολίες. Από τεχνικής πλευράς λοιπόν δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε την ε, τεχνολογική ουδετερότητα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να προωθούμε πληροφορίες ε, κατά τρόπον ώστε ε, τα άτομα που έχουν αναπηρίες να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ε, πληροφορίες. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο ε, λογισμικό, το οποίο να είναι ένα καθολικό λογισμικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καπάτο και τώρα ο κύριος Σάση από το Φιλανδικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Φιλανδικό Κοινοβούλιο έχει επίσης ορισμένες αμφιβολίες ως προς τον προτινόμενο κανονισμό εμείς θεωρούμε ότι η δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα λειτουργεί πολύ καλά μέχρι τώρα. Από τότε που πρώτο άρχισε να εφαρμόζεται ο κανόνας της διαφάνειας το 2001 και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε αυτό, ακριβώ αποφάσισε και πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του. Ο κύριος Κάσμαν υπήρξε πολύ δραστήριος και νομίζω ότι η προσέγγιση του είναι σωστή. Θα ήθελα όμως να θέσω και δύο ερωτήματα. Πρώτον, όσον αφορά την έννοια του εγγράφου, δεν κατάλαβα ακριβώς τις ανησυχίες της κυρίας Γουάλτρομ. Μπορεί να μας πει σαφέστερα ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Κομισιόν και τα άλλα όργανα της Ένωσης για να ανταποκριθούν στα αιτήματα για χορήγηση εγγράφων. Μήπως δεν υπάρχουν αυτά τα έγγραφα, ποια είναι η δικαιολόγηση των αρνήσεων. Ξέρω ότι μπορεί να υπάρχουν και τεχνικοί φραγμοί, αλλά να μου τους πείτε. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει συνένεση ότι είναι προβληματική η κατάσταση και ότι χρειάζεται βελτίωση. Παραδείγματο χάρη να αναφερθήκατε στη σύσταση που έκανε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για την καταχώρηση των εγγράφων, αλλά από ό,τι ξέρω όλα τα έγγραφα που υπάρχουν είναι κατακεχωρημένα. Αλλά από ό,τι ξέρω ακόμη και τα μη καταχωρημένα έγγραφα μπορείτε να τα διαθέσετε. Το σύστημα λοιπόν δεν νομίζω ότι χρειάζεται βελτίωση. Μπορείτε λοιπόν επαναλαμβάνω να μας ξαναπείτε γιατί δεν αρκεί ο υπάρχον ορισμός. Δεύτερο ερώτημα προς τον κύριο Κάσμαν. Τα έγγραφα που προέρχονται από τις χώρες μέλη είπατε ότι θέλετε να δοθεί δικαίωμα βέτο στα κράτη-μέλη ώστε να μην μπορεί να, δοθεί, να χορηγηθούν ορισμένα έγγραφα που έχουν υποβάλει στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Πώς συμβαδίζει αυτό με τον κανόνα της διαφάνειας. Εάν αυτό το δικαίωμα του βέτο δεν γίνει δεκτό, μήπως έτσι θα υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Αυτό αναρωτιέμαι. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μοντενέγκρο. Μόνο δύο λεπτά όμως τον παρακαλώ γιατί περιμένουμε και τις απαντήσεις του αντιπροθυπουργού μας που πρέπει να φύγει σε λίγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Εντάχει θα θέλαμε να πούμε και εμείς ε, τη γνώμη μας. Σε σχέση με τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ύψης της σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για θέματα ευρωπαϊκής ηθαγένειας που μας απασχόλησαν χτες. Είναι αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας και αποτελεί βεβαίως είναι η, η, η κορονίδα της πρόσβασης στα έγγραφα και αφορά και την ίδια τη δημοκρατική μας νομιμότητα. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ηθαγένεια αν δεν υπάρχει λογοδοσία από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ε, δυστυχώς υπάρχουν περιορισμοί όταν υπάρχουν θέματα δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και βεβαίως υπάρχει και το ε, απόρριτο των επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Εμείς στην Πορτογαλία έχουμε ένα σύστημα πρόσβασης που λειτουργεί πολύ καλά. Υπάρχει μια κοινοβουλευτική επιτροπή που κάνει μια πρώτη διαλογή των αιτήσεων πρόσβασης από πλευράς ε, πολιτών ή δημόσιων διοικήσεων, δημόσιας διοίκησης, όταν έχει ορισμένες αμφιβολίες και θα ήθελα να πω ότι το 95% των αιτήσεων κοινοποιείται. Και ε, με βάση αυτό το αρχικό κοσκίνισμα που σας είπα, όλα ε, βρίσκονται Μάλλον σε όλα έχει πρόσβαση το κοινό και οι πολίτες. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να άρουμε αυτά, αυτές, αυτούς τους διχασμούς που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, ε, Ευρω, ε, Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού καθώς και Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει ιδιαίτερα αυτό το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και πολιτών. Εάν οπισθοχωρήσουμε, τότε στην ουσία ε, πολεμούμε και καταπολεμούμε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Τώρα ήρθε η ώρα να παρέμβει ο κύριο Σάσα Βόντρα. Σα ευχαριστώ πολύ για τα ε, σχόλιά σας και ευχαριστώ και για την πρωτοβουλία που πήρατε ε, να κάνετε τόσο νωρίς αυτή τη συνεδρίαση για να σηματοδοτηθεί η έναρξη της Προεδρίας. Ευχαριστώ την κυρία Βάστρομ, ευχαριστώ τον Μάικλ Κάσμαν για τη σκληρή δουλειά του σε αυτό τον τομέα κάνει μια σοβαρή ανάλυση του προβλήματος. Όλοι καταλαβαίνουμε τις παραμονές και των εκλογών στο Κοινοβούλιο, ε, πόση σημασία έχει αυτό το θέμα της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα και η διαφάνεια πόσο σημαντική είναι για να ε, αυξηθεί η συνθητοποίηση του κόσμου. Είναι ένα θέμα και πολιτικής έτσι, διάστασης. Άκουσα τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Στην περίπτωση του κυρίου Τούρκο, στην απόφαση, δεν ε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει από το καλοκαίρι του 2008 η απόφαση του ΔΕΚ βέβαια. Δεν ξέρω αν ελήφθησαν, λέτε, τα απαραίτητα μέτρα από το Συμβούλιο. Ορισμένες νομικές νομοδοτήσεις όντως ε, ε δεν δόθηκαν λόγω της ευαίσθητης φύσης τους, αρνήθηκαν την πρόσφασή τους. Αλλά γενικά το Συμβούλιο αντέδρασε θετικά. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή, είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει όλοι να τη συνοψίσουμε ως εξής. Θα συνεχιστεί η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσβλέπουμε ε, στην τελική έκθεση που θα πρέπει να συμπεριληφθεί ε, στις εργασίες της Επιτροπής Ελευθεριών και αν δεν απατώμε ε, περί τα μέσα Φεβρουαρίου θα ψηφιστεί στην Επιτροπή θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα ότι υπάρχει ένα καθεστώς πρόσβασης στα έγγραφα σήμερα το οποίο εφαρμόζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαρακτηρίζεται ακριβώς από μια ροή πληροφοριών. Υπάρχουν σημαντικά χαρακτηριστικά δεδομένα. Πρώτον, η ύπαρξη γενικής πρόσβαση. Ε, αναγνωρίζεται το γενικό δικαίωμα των πολιτών στην πρόσβαση. Ε, πολύ ευρεία επίσης ε, ε, η έννοια του εγγράφου και του ορισμού. Στη συνέχεια θα πρέπει κάθε θεσμικό όργανο να ε, εξετάζει βέβαια περίπτωση τα έγγραφα που ζητεί το κοινό βάσει της λεγόμενης ε, δοκιμής ζημίας, δηλαδή ποια είναι η πιθανή ζημία που μπορεί να προκληθεί για το θεσμικό όργανο η δημοσίευση του εγγράφου αυτού. Και ένα τελευταίο, χωρίς να είναι αυτό το λιγότερο σημαντικό, η ύπαρξη ε, διοικητικών ή νομικών επιφυλάξεων κατά των αποφάσεων ε, ή μάλλον υπάρχει δυνατότητα διοικητικής ή νομικής προσβηγής και δικαστικής ακόμα. Ε, υπάρχει λοιπόν ο κανονισμός 1049 του 2001 που δεν θα πρέπει να διακυβευτεί και να υπονομευθεί διότι λειτουργεί σωστά. Θα πρέπει να εδραιωθεί λοιπόν αυτό το κεκτημένο, να κατοχυρωθεί βρίσκοντας το σωστό ε, μέσο όρο, τη χρυσή τομή ανάμεσα στα δικαιώματα των πολιτών για την πρόσβαση του έγγραφα και την προστασία κάποιας ε, μορφής ιδιωτικών και δημοσίων συμφερόντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ε, ε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, καλή σας πτήση και καλή σας προσγείωση. <laughs> Πρωτίστως, λέει ο μιλητής. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μάργο του τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνεισφορά όλων. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή σε σχέση με τον ολοκληρωτικό απολογισμό του κανονισμού 1049 τα τελευταία 7 χρόνια και γι' αυτό ζητήσαμε μία αναθεώρηση, ένα recast για να δούμε ποιες είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις, να ευθυγραμμιστούμε με τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Παράλληλα, αυτή η συζήτηση αντικατοπτρίζει τα συγκρόμενα συμφέροντα που υπάρχουν ορισμένες φορές. Προσπαθούμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο δυνατό πεδίο, γιατί μιλάμε για την πρόσβαση του κοινού στην ε, πληροφορία και θέλουμε να καλύψουμε να καλύψουμε πραγματικά ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος ε, του κενού που υπήρχε μέχρι τώρα. Βλέπουμε και τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τη χρήση των ε, στοιχείων από το κοινό και ε, πάνω από 70% των αιτήσεων προέρχονται και αφορούν ευρωπαϊκές υποθέσεις. Δηλαδή, κάτω από 30% αφορά γενικά το κοινό και ούτε οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν αυτό το δικαίωμα εκτεταμένα. Και βεβαίως υπάρχει και ενδιαφέρον από τον ακαδημαϊκό κόσμο και πρωτίστως όπως σας είπα από τη δημόσια διοίκηση 70%. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε το ευρύτερο δυνατό πεδίο και παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει νομική διαφάνεια γιατί δεν έχει νόημα να υπάρχει ασάφεια, μεγάλη ασάφεια γιατί τελικά δεν ε, λαμβάνουμε πληροφορίες, αλλά πληθώρα χαρτιών και τίποτα άλλο. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε και να προωθήσουμε και το δικαίωμα πρόσβασης. Όσο πιο ασαφής ε, είναι κανείς, τότε πιο, τόσο και πιο αυθαίρετο θα είναι για τα θεσμικά όργανα να κρίνουν τι θεωρείτε εσείς ως έγγραφο. Γι' αυτό μπορεί ένα θεσμικό όργανο να θεωρήσει ότι ένα στοιχείο αποτελεί έγγραφο, ένα άλλο όχι. Αυτό είναι ένα εγγενές ζήτημα. Άρα αν υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, τόσο το καλύτερο. Για να έχετε τη σωστή πρόσβαση. Επίσης ε, θέλουμε να υπάρχει ένα ανοιχτό πεδίο και μεγαλύτερη διαφάνεια καθώς και πρόσβαση. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα, με ιδιωτικά στοιχεία ή με τον χώρο περισυλλογής των διαφόρων πολιτικών φορέων. Δηλαδή υπάρχει ένας ορισμός που στο τέλος οι βουλευτές δεν έχουν χώρο για να μπορέσουν να διαβουλευτούν ή να σκεφτούν ένα ζήτημα σωστά. Άρα δεν τους έχετε βοηθήσει. Αυτή είναι μια δυναμική των θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό και στο σουηδικό σύστημα, το οποίο είναι το πλέον ανοιχτό και διαφανές, Πολλές φορές ορίζουμε ένα έγγραφο ως ε, έγγραφο εργασίας, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό. Και υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις και στο σουηδικό σύστημα για να μπορέσει να είναι λειτουργικό. Γι' αυτό μας ενδιαφέρουν οι ορισμοί πρωταρχικά. Και απορρίπτω την ιδέα της ε, λιγότερης πρόσβασης. Θέλουμε να είναι μεγαλύτερη η πρόσβαση και αυτό ήταν το σημείο εκκίνησης της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε μεγαλύτερη πρόσβαση. και βεβαίως ευρύτερο ορισμό για το ποιος έχει πρόσβαση, δηλαδή όχι μόνο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ε, τον υπολογιστή του και δεν ξέρουμε ε, γιατί χρησιμοποιεί κανείς τα στοιχεία. Ναι. Γι' αυτό θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις ε, τεχνολογικές αλλαγές και θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε και την νομοθεσία υπ' αυτή την έννοια. Επίσης, σας ανέφερα ότι υπάρχουν ενδιαφέροντες τρόποι ε, διατύπωσης για να είμαστε σαφέστεροι για το τι θέλουμε να επιτύχουμε. Δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση και μεγαλύτερη διαφάνεια. Και αν βρούμε τις κατάλληλες λέξεις θα τις δεχτούμε. Η συζήτηση δείχνει ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία και διατυπώσεις οι οποίες στην ε, εφεξής διαδικασία θα μας απασχολήσουν. Και το και ή ίσως είναι καλύτερο από το να υπάρχει και σε ένα σημείο και ή διαζευκτικό σε ένα άλλο. Αυτό το είδαμε και στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και θα το δούμε και στην μελλοντική διαδικασία. Επίσης, ακούω τις φιλοδοξίες, ε, ο κύριος Κάσμαν την εξέφρασε αυτή τη φιλοδοξία. Δεν μπορούμε όλα να τα εντάξουμε στον 1049. Θα πρέπει να ξέρουμε τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή πού στοχεύει αυτός ο κανονισμός και μετά θα έχουμε, θα προωθήσουμε συμπληρωματικές προσπάθειες βεβαίως. Έχουμε ένα σύστημα καταχώρησης στην Επιτροπή. Αυτό όμως δεν ισχύει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στα άλλα θεσμικά. Άρα δεν υπάρχει απλός τρόπος επίλυσης. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει ευθυγράμμιση και εναρμόνιση για να έχουμε ίδιο τρόπο εφαρμογής και καταχώρησης. Και αυτό αφορά συμφωνίες μεταξύ θεσμικών οργάνων. Σε μερικές περιπτώσεις, πολλοί ζήτησαν μεγαλύτερη εμβέλεια και αυτό σημαίνει ότι αν ε, η νομοθεσία δεν καλύπτει τα ίδια στοιχεία, τότε δεν είναι αποτελεσματικό ε, να πούμε ότι θα γίνει διεύρυνση ή κάτι θα αρχιοθετηθεί ή όχι. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο του 1049. Θα γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές εάν κάποια στιγμή εφαρμοστεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου, ότι θα μας βοηθήσει και θα διευρύνει την, την εμβέλεια του κανονισμού. Κύριε Καπάτο, αυτό δεν είναι υπηρεσία στους πολίτες, είναι δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να είμαστε πραγματιστές και στην Επιτροπή. Εάν Υπάρχουν πολλά λόμπι, οι ε, δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες κρίνουν ότι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα έγγραφο, σε μία έρευνα η οποία διενεργείται μία συγκεκριμένη στιγμή, θα πρέπει να μπορέσουμε να ελέγχουμε όλες τις σελίδες κάθε εγγράφου και άρα στο τέλος δεν θα είναι προσβάσιμο. Πρέπει όμως να το κάνουμε αυτό ή πολλές φορές πρέπει να αφαιρέσουμε ονόματα από συγκεκριμένα έγγραφα. Για να υπάρχει λοιπόν νομική ασφάλεια, νομική διαφάνεια, θα πρέπει να πούμε ότι για έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό ή όχι. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση ή όχι. Έτσι μπορούμε να προωθήσουμε την ε, διάδοση, την πραγματική διάδοση των εγγράφων, παρά να χάνονται τα χρήματα των φορολογούμενων άσκοπα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Έτσι λειτουργήσε το σύστημα μέχρι τώρα. Αυτά είναι μερικά στοιχεία που όφυλα να υπογραμμίσω Θέλουμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση στα έγγραφα, όλοι το επιθυμούμε αυτό. Φέρουμε συγκεκριμένη ευθύνη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από τον κανονισμό, δηλαδή πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον κανονισμό έτσι ώστε να εξυγχρονιστεί και να λάβει υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του 10 στην περίπτωση Τούρκο και άλλες υποθέσεις. Τώρα υπάρχει κάλυψη και θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το πλαίσιο έτσι ώστε να ακολουθούμε τις αποφάσεις του ΔΕΚ. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μελλοντικά για τη βελτίωση της πρόσβασης στα έγγραφα. Ευχαριστώ. Πολύ κυρία Αντιπρόεδρέ μου και τώρα θα δώσω το λόγο στον τελευταίο μιλητή, τον Μιχαήλ Κάσμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι συντομότατος. Είναι Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση και αυτά που μας είπε η Αντιπρόεδρος Βάλστρομ, γιατί ο καθένας ακούει μια συζήτηση και παίρνει από αυτήν αυτό που τον ενδιαφέρει. Εγώ αυτό που άκουσα είναι ότι οι προτάσεις από την Κομισιόν είναι η παναχώρηση. Αυτό ακούστηκε ως κριτική και το είπαν και πολλοί εθνικοί βουλευτές. Ξέρω ότι είναι σωστή και καλή πρόθεση της Κομισιόν και βασίζεται στην επταετή εμπειρία που είχαμε από την εφαρμογή του κανονισμού. Αλλά η κυρία Βάλστρομ ασχολείται με τα θέματα της διαφάνειας πολύ περισσότερο χρόνο από μένα και εγώ έχω φτάσει να ενδιαφερθώ σε αυτό το θέμα από την άποψη του αστυνομικού Δηλαδή, ποια κατάχρηση θα μπορούσε να γίνει της νομοθεσίας αυτής. Και γι' αυτό οι τροπολογίες μου στοχεύουν στην αποτροπή της κατάχρησης, στην παρεμπόδιση της κατάχρησης. Γι' αυτό μιλήσαμε για νέο ορισμό. Αν κάποιος δεν έχει υποβάλει επίσημα κάποιο έγγραφο, δεν θεωρείται έγγραφο αυτή τη στιγμή ενώ θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η Κομισιόν δεν συμφωνεί βέβαια μαζί μου, αλλά αυτό σημαίνει απλώς ότι η συζήτηση θα είναι πιο ενδιαφέρουσα. Επίσης, μου άρεσε η άποψη ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε αντιτιθέμενα συμφέροντα. Αλλά αυτό ακριβώς είχε κάνει η πρόταση του 2001. Πρέπει απλώς να δούμε προς τα που πρέπει θέλουμε να προχωρήσουμε ας πούμε όταν λήξει μία έρευνα να υποβάλλονται τα έγγραφα μετά το τέλος της έρευνας διότι η καλή διακυβέρνηση είναι κάτι το πολύ ουσιώδες για την καλή λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Αν με παίρνει κανείς τηλέφωνο, παρακαλώ λέω στο βοηθό μου πες του ότι θα πάρω αργότερα, δεν θέλω διαφάνεια και σε αυτά. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε πράγματα που δεν μπορούμε να τα αναστρέψουμε. Δεν υπάρχουν προνόμια και εξαιρέσει από την διαφάνεια. Η εξυπηρέτηση των πολιτών μας είναι τιμή μας. Θεσμικά θα διευκολύναμε πάρα πολύ τα πράγματα αν υπήρχε ένας ειδικό αξιωματούχος για την πληροφόρηση, αν ήταν διαθέσιμα όλα τα έγγραφα καταχωρημένα και υπήρχαν σαφέστατοι κανόνες μόνο για τις εξαιρέσεις, όταν δεν πρέπει να καταχωρηθεί κάποιο έγγραφο δηλαδή. Ο Ισπανός συνάδελφος μίλησε για ισότητα της πρόσβασης. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα. Πώς είναι δυνατόν να διασφαλιστεί το δικαίωμα της πρόσβασης σε αυτά που αφορούν τον ίδιο τον πολίτη. Αρνούμε λοιπόν τα προνομιακά δικαιώματα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ιεραρχημένη πρόσβαση. Ορισμένοι δημοσιογράφοι μου το ζήτησαν, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν δίκιο. Εγώ θα ήθελα να διασφαλίσω ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν ίση μεταχείριση. Έχουμε ξαναμιλήσει για το θέμα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αλλά δικαιοσύνη σημαίνει λογοδοσία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπουργοί πρέπει να προστατευτούν στην ιδιωτική του ζωή αλλά η διαφάνεια σημαίνει ότι πρέπει ορισμένα ουδέτερα προσωπικά στοιχεία να χορηγούνται ως θέμα αρχής για την διαφάνεια να προστατευθεί ο χώρος της ιδιωτικής καθαρά σκέψης αλλά να υπάρχει πρόσβαση ακόμη και στις πιο περίεργες και ακραίες ιδέες. Ιδέες είναι που μπορούν να συζητηθούν. Δύο τελευταία. Η Λισαβόνα βέβαια τα αλλάζει όλα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να εργαστούμε πολύ αποτελεσματικά όταν και αν επικυρωθεί. Στην Ιρλανδία, η Ιρλανδία πέριψαν εν μέρη γιατί θεώρησαν ότι δεν έτυχαν καλής πληροφόρησης. Και έρχομαι λοιπόν στο ερώτημα που έθεσε ο κύριος Σάση από τη Φιλανδία. Στην τροπολογία μου προς το άρθρο 5.2 αναγνωρίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη θέλησαν να μην υπάρχει πρόσβαση σε έγγραφα που είχαν υποβάλει. Εγώ θα ήθελα να δοθεί μια βάση σε τέτοιες διαδικασίες στην ίδια τη συνθήκη στο 296 για τις, τους όρους με τους οποίους ένα έγγραφο μπορεί να μην χορηγηθεί. Και για να επανέλθω στο Σέξπιρ, το Σάντσο Πάνσα και το Δον Κιχώτη θα παραφράσω κάτι από το τέλος του βασιλιά Λίρ όπου υπάρχει μια κατάχρηση εξουσίας και πόλεμος πριγκίπων με πρίγκιπες. Παραφράζω για να μην αναφερθώ στον πονηρό που λέει το πρωτότυπο. Λέει ο Σέξπιρ το κακό που διαπράττουν οι άνθρωποι διατηρείται αλλά το κακό θάβεται μαζί με το σώμα τους. Το 1049 λοιπόν του 2001 δεν είναι δυνατόν να το θεωρήσουμε κακό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί η τέταρτη συζήτηση θα καθυστερήσει. Λοιπόν, Μπορεί να μακρηγορήσαμε, αλλά νομίζω ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και θα δούμε τι συμπεράσματα θα βγουν και τον επόμενο μήνα. Ο επόμενος, ο πρόεδρος της επόμενης συζήτησης είναι ο κύριος Ζεράρ Ντεπρέ.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 αλλά δεν πειράζει γιατί ήταν πραγματικά συναρπαστική η συζήτηση. Περνούμε λίγο στην τελευταία ενότητα που εγγράφεται στη συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης και τη διευρύνει και τη συζήτηση και την αντιπαράθεση που είχαμε. Ε, βάσει και πέρα από την πρόσβαση στα έγγραφα, Ασχολείται την ενότητα αυτή με τη βελτίωση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω σωστά θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να αποτανθούμε σε εκπροσώπους κρατών που έχουν μη τι άλλο τη φήμη αλλά και την ε, εμπειρία και την πρακτική καλών ε, συνηθιών για τη διαφάνεια και την πρόσβαση στα έγγραφα. Η διαφάνεια κατά τη διαδικασία αποφάσεων είναι πραγματικά επιταγή. Επιβάλλεται δηλαδή όχι μόνο στα θεσμικά όργανα της Ένωσης αυτά καθ' αυτά, αλλά και στο σύνολο των κρατών μας. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα όλων των θεσμικών οργάνων. Ε, βάσει αυτών όλων λοιπόν των βέλτιστων πρακτικών, έχει σημασία και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπνευστούν από τα όσα θα ακούσουμε σήμερα. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Υπουργό, την κυρία Μπέατρης Άσκ, Υπουργό Δικαιοσύνης ε, του Βασιλείου της Σουηδίας. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω ότι αποτελεί για μένα τιμή η πρόσκληση που μου απευθύνεται και η δυνατότητα, η ευκαιρία που είχα να ε, παρακολουθήσω την προηγούμενη συζήτηση. Πιστεύω γενικά ότι η διαφάνεια γενικά και ειδικότερα η πρόσβαση στα έγγραφα προάγει τη ε, δημοκρατία, επιτρέπει στους πολίτες να ασκήσουν έλεγχο ε, στην εξουσία και στη διοίκηση και βοηθάει στην αποτελεσματικότητα ε, της δίκησης και καταπολεμά τη διαφθορά. Και τελικά δεν είναι μεγαλύτερη νομιμότητα σε κάθε κυβέρνηση. Πρώτα μου στήθηκε να μιλήσω για τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη-μέλη. Στη δική μου περίπτωση πρόκειται για τη Σουηδία και το δικαίωμα πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα είναι ακρογωνίως λήθος ε, του συντάγματος και της νομοθεσίας μας. από τον 18ο ε, αιώνα και εγώ ως υπουργό Δικαιοσύνης είμαι αρμόδια για αυτά τα θέματα και για άλλα θέματα πρόσβασης ε, στη νομοθεσία και θα ξεκινήσω από εδώ. Θα επικεντρωθώ σε μερικές γενικές αρχές που είναι ενδιαφέρον να συζητήσουμε υπό το φως της αναθεώρησης του κανονισμού για την πρόσβαση του κοινού στα κοινοτικά έγγραφα. Ε, το Σύνταγμα της χώρας μου δίνει το δικαίωμα πρόσβαση στους πολίτες κάθε γράφου που καταρτίζει ή ε, ε, εκδίδει ε, κάποια κρατική αρχή σε οποιοδήποτε μέσο, σε οποιαδήποτε πληροφορία, καλύπτονται όλα τα υποστρώματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα τα έγγραφα ναι. είναι πλήρως προσβάσιμα. Στο Σύνταγμα επίσης αναγράφεται ένας κατάλογος εξαντλητικός ιδιωτικών και δημοσίων συμφερόντων που θα πρέπει να διαφυλάσσονται και να προστατεύονται. Υπάρχει νόμος περί απορρίτου πάρα πολύ ε, αναλυτικός για ευαίσθητα ε, έγγραφα όπου αρνείται η δημοσίευση, ε, τη δημοσίευσή του στο δημόσιο. Πάντα κάθε αίτημα θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και με κάθε ευκαιρία να αξιολογούνται τα αιτήματα. Έχουμε λοιπόν κανόνες που συνδέονται με όλα τα έγγραφα σας είπα των δημοσίων αρχών έχουν πρόσβαση πολίτες εκτός αν υπάρχει εξαίρεση ε, περί απορρίτου σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Σύνταγμα. Και είναι αρκετά εύκολο για τον απλό πολίτη να έχει πρόσβαση. Η διοίκηση, η κυβέρνησή μας ε, είναι συνηθισμένη να χειρίζεται τα θέματα αυτά και είναι πάρα πολύ σπάνιο να ακούει κανείς παράπονα ή καταγγελίες. Ε, από πλευρά της διοίκησης δηλαδή ότι είναι υπερβολική η καταγγελιες απο πλευρα τη διοικηση δηλαδη ή δεν μπορεί να δοθεί συνέχεια. Ε, το ευρωπαϊκό σύστημα έχει πολλές αντιστοιχίες στα χαρακτηριστικά του. Σήμερα όλα τα έγγραφα είναι δημόσια ε, των τριών θεσμικών οργάνων, εκτός αν άλλος ορίζει ρητά ο κανονισμό περί απορρίτου. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές με το σουηδικό σύστημα. Η βασική διαφορά είναι ότι μόνο τα τρία θεσμικά όργανα και όχι όλα τα όργανα της Ένωσης ε, καλύπτονται από αυτή τη ρυθμίση. Ενώ στη Σουηδία αυτό αφορά όλα τα κρατικά όργανα και όλες τις δημόσιες αρχές και έχουν το δικαίωμα οι πολίτες να τα συμβουλεύονται. Θα πρέπει πάντα να βρούμε την ισορροπία μεταξύ του θεμελιωδούς δικαιώματος αλλά και ε, την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών. Πάνω από 200 χρόνια εμείς εφαρμόζουμε αυτό το συνταγματικό δικαίωμα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις από το 2001 και μετά. Θα ευχόμαστε και η Ευρώπη να λειτουργεί όπως η Σουηδία. Μα ρωτώ, με χρειάζεται να αλλάξει το συγκεκριμένο τόσο νωρίς μετά την έγκριση του κανονισμού του 2001. Γιατί τόσο σύντομα. Άκουσα την προηγούμενη συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κάτι για τον κανονισμό που γνωρίζετε και δεν χρειάζεται να σας επαναλάβω την πρόταση. Υπάρχουν όμως ε, ερωτηματικά και ανησυχίες και αφορούν και τη συζήτηση στο εσωτερικό της Σουηδίας. Πρώτον, τι εστί έγγραφο, ε, με βάση ποια κριτήρια. Δεν άκουσα κανένα πρακτικό πρόγραμμα πουθενά μέχρι τώρα στη Σουηδία να γνωρίζω τι είναι έγγραφο. Δεν άκουσα τη συζήτηση δεν, δεν άκουσα ποτέ κανένα που να λέει ότι είναι πολύ ασαφής η έννοια για να χρησιμοποιηθεί και να ε, εφαρμοστεί στην πράξη. Όταν επίσης ε, υπάρχει πρόταση να αποκλείονται ορισμένε κατηγορίε εγγράφων, εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν εξαιρεσει ήδη για έρευνε που διεξάγονται Και δεν χρειάζεται να αλλάξει μια αρχή τέτοια με βάση κάποια απόφαση ενό μεμονωμένου πολίτη. Εν πάση περιπτώσει δεν με αφορά αυτό το θέμα. Ε, στη συνέχεια υπάρχει εξή κίνδυνο. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ένωση είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει πάρα πολύ τη διαφάνεια. Υπάρχει μάλλον κίνδυνος να έχουμε το αντίστροφο αποτέλεσμα επιπλέον και θα επανέλθω στη συνέχεια, θα είναι πολύ πιο δύσκολο ο κόσμος να καταλάβει αυτούς τους κανόνες. Και θα πρέπει εμείς εδώ ξεκάθαρα να λέμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι πολίτες. Αυτοί θέλουν τις πληροφορίες και αυτούς θα πρέπει να διευκολύνουμε. Δηλαδή ακόμα και αν είναι δικηγόροι, εταιρείε, η τελική ανάλυση άνθρωποι είναι αυτοί που ζητούν τις πληροφορίες. Γιατί θέλετε να εξαιρούνται αυτές οι ομάδες, οι δικηγόροι, τα λόμπι, πάντα άνθρωποι δεν είναι κι αυτοί. Τώρα αν είναι πιστοδρόμης ή ή πρόοδος, δεν ξέρω. Αν μπούμε σε αυτό το έδαφος είναι πολύ αληστηρό. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να πάμε στην άλλη κατεύθυνση και να το παρακάνουμε ε, από την πολύ διαφάνεια. Γιατί πέρα από τη διαφάνεια, αυτό που μα ενδιαφέρει είναι σαφή και η γλώσσα μα. Δηλαδή, ο στόχο είναι να καταλαβαίνει ο κόσμο αυτό που είναι γραμμένο στην νομοθεσία και στο οποίο έχει πρόσβαση. Όπω μπορεί να γνωρίζετε, δεν είναι εύκολο καμιά φορά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύσκολο να διαβάζει κανεί τα όργανα. Πέρα από την νομοθεσία, θα πρέπει να δουλεύουμε λοιπόν και στη διατύπωση. Και, κατά τη διάρκεια τη Σουηδική Προεδρία θα γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο σχετικά. Γιατί είναι ο ίδιο στόχο Θα πρέπει οι πολίτες λοιπόν να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται και να καταλαβαίνουν το έγγραφο που διαβάζουν όταν θα αποκτήσουν την πρόσβαση σε αυτά. Βέβαια υπάρχουν τα θέματα της νομιμότητας, της εμπιστοσύνης που σας ανέφερα στην αρχή. Για τους πολιτικούς είναι προφανές ότι έχει μεγάλη σημασία να μας εμπιστεύεται ο κόσμος. Πολλοί θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση μυστική λέσχη. Θα ήθελα να σας το πω εδώ, γνωρίζουμε όλοι ότι βλέπουμε ανθρώπους, καθημερινούς πολίτες στον δρόμο που θεωρούν ότι είναι δύσκολο να ενημερωθούν και επίσης θεωρούν ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι ίδιοι ε, στη νομοθετική δουλειά, ότι είναι αποκλεισμένοι από αυτή. Εγώ θέλω οι πολίτες να θεωρούν ότι είναι ενεργοί ε, φορείς, πρωταγωνιστές του γίγνεσθε στην Ευρώπη. Ε, θα ε, ήθελα να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό επανερχόμενη στη Σουηδία. Να είναι πραγματικό ε, δικαίωμα για όλους τους πολίτες. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η καταχώρηση, η πρωτο, πρωτοκόλληση όλων των εγγράφων που καταρτίζονται ή λαμβάνονται, παραλαμβάνονται από κάποια δημόσια αρχή θα πρέπει να πρωτοκολούνται. Για να δούμε αν είναι ένα έγγραφο που ενδιαφέρει το πολίτη ουσιαστικό. Βέβαια αυτή η καταχώρηση είναι πολύ σημαντική ε, για να πιστοποιεί την ε, ύπαρξη καν ενός εγγράφου, αλλά θα πρέπει να έχει τη διαδικασία, τη δυνατότητα, συγγνώμη, ο πολίτης να συμβουλεύεται αυτό το μητρό. Και αυτό είναι δημόσιο στη Σουηδία. Βεβαίως υπάρχει χώρος ε, βελτίωση. Στα Σουηδικά Μητρώα θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη νομοθεσία και κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και κατάρτιση του προσωπικού για να μπορούν όλοι να χειρίζονται σωστά αυτά τα ε, μητρώα. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα ευρύ κατάλογο και μητρό ή περισσότερο. Και εκεί πραγματικά ψάχνουν οι απλοί πολίτες ε, σε αυτά τα μητρώα, γιατί οι υπόλοιποι ξέρουν που θα τα βρουν μάλλον. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας ε, παρουσιάσω τις απόψεις μου. Ε, ευχαριστούμε πολύ κυρία μου, κυρία Υπουργέ, για την ενδιαφέρουσα αυτή εισήγηση. Εγώ αμέσως βλέπω τι σημαίνουν όλα αυτά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα η έννοια clear language. Νομίζω ότι είναι θέμα επί του οποίου πρέπει να κάνουμε ακόμη πολλές προσπάθειες στην επόμενη θητεία. Λοιπόν, ας μην μακρηγορήσω, θα δώσω αμέσως το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμικών Θεμάτων της Φιλανδικής Βουλής, τον κύριο Κίμο Σάση. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι κυρίες και κύριοι, Χωρίς μικρόφωνο. Κυρίε και κύριοι, σα είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για τη διαφάνεια στη Φιλανδία. Χαίρομαι επίση ιδιαίτερα γιατί οι οργανωτέ διάλεξαν τη Φιλανδία ω εκπρόσωπο τη περισσότερο διαφανούς χώρας μέλου μαζί με τη Σουηδία. Το 89 όταν, ήταν, ε, όταν η Φιλανδική Προεδρία από τις πρώτες, 90 είναι, από τις πρώτες μας προτεραιότητες ήταν η διαφάνεια. Και εγκρίθηκε το 2001 επί για μένα είναι μεγάλη ευχαρίστηση που μιλώ μετά τον Υπουργό Δικαιοσύνη τη Σουηδία και αυτό με διευκολύνει ιδιαίτερα γιατί η διαφάνεια των δημοσίων δραστηριοτήτων είναι μεγάλη προτεραιότητα και τη Σουηδία και τη Φιλανδία, τουλάχιστον από το 1766 όταν πέρασε το πρώτο νομοσχέδιο για την ελευθερία τη πληροφόρηση. Η Φιλανδία εκείνη την εποχή ήταν τμήμα του Βασιλείου τη Σουηδία. Ε, γι' αυτό έχουμε την ίδια βάση στην νομοθεσία μα. Θα ήθελα απλώ να αναφέρω ότι ο Άντερ Κιντένιου ένας Φιλανδός παπάς και μέλος του Συνδικού Κοινοβουλίου θεωρείται ο πατέρας του νομοσχεδίου εκείνου. Και το προήμιο του νομοσχεδίου αυτού που έχει ηλικία 250 ετών λέει αφού σκεφτήκαμε τα μεγάλα θετικά στοιχεία που υπάρχουν για την πληροφόρηση του κοινού και του τύπου και επειδή η αμοιβαία πληροφόρησε διάφορα χρήσιμα θέματα, προωθεί την ανάπτυξη και διάδοση των επιστημών και των τεχνών, αλλά επίσης δίνει μεγαλύτερες ευκαιρίες σε όλους μας τους υπηκόους να μάθουν κάτι παραπάνω και να μπορούν να κρίνουν για την καλύτερη τους διαχείριση αποσιοποιητικά. Και μετά λέει το νομοσχέδιο ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και να λαμβάνει εγκεκριμένα αντίγραφά τους. Ήδη από το 1766 υπήρχε μάλιστα και κύρωση που προβλεπόταν αν δεν χορηγούνταν η ετούμενη πληροφορία. Εγώ δεν προτείνω κυρώσεις εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον όχι αμέσως. Αλλά ε, η κύρωση αυτή ήταν πολύ αποτελεσματική. Λοιπόν, μαζί με τη Σουηδία έχουμε παρόμοια συστήματα που βασίζονται στην ίδια ιδέα της διαφάνειας που θα μπορούσε κανείς να την ονομάσει βόρειο πρότυπο. Ο στόχος είναι άτομα και ομάδες ατόμων πολιτών να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους για την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Αυτό τους επιτρέπει να κρίνουν σωστότερα και να συμμετέχουν καλύτερα στη δημόσια συζήτηση για να επηρεάσουν τη διαχείριση κοινών θεμάτων και επίσης ενδυναμώνει το δημοκρατικό χαρακτήρα και την ομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ενδυνισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού. Δείτε στη Σουηδία πόσο καλά πήγαν όλα με αυτό το θέμα της διαφάνειας δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα. Στη Φιλανδία το δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα είναι βασικό δικαίωμα που προστατεύεται από το Σύνταγμα. Σύμφωνα με το τμήμα 12 του Συντάγματος, όλα τα έγγραφα που κατέχουν οι δημόσιες αρχές είναι δημόσια, εκτός εάν για δικαιολογημένους λόγους υπάρχει περιορισμός. Αυτή η ρήτρα εκφράζει την αρχή της διαφάνειας που βασίζεται στην πεποίθηση ότι η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα είναι ο κανόνας και ο περιορισμός η εξαίρεση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει απαγόρευση χωρίς σαφή δικαιολόγηση και αναφορά των συμφερόντων που προστατεύονται από την απαγόρευση. Εκτός αυτού το Σύνταγμα και η Συνταγματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου της Φιλανδίας έχει τονίσει επανειλημμένος ότι οι περιορισμοί στη διαφάνεια πρέπει να ερμηνεύονται στενά. Παραδείγματο χάρη ότι το copyright ακόμη και για τα επίσημα έγγραφα μπορεί να είναι απαράδεκτος περιορισμός της δημόσιας συζήτησης και της ελεύθερης διακίνησης της πληροφόρησης. Το νομοσχέδιο που εφαρμόζεται σήμερα λέγεται νομοσχέδιο για την διαφάνεια των κυβερνητικών δραστηριοτήτων και ενεκρίθη το 1999. Το εύρος του είναι πολύ μεγάλο γιατί καλύπτει όλες τις δημόσιες αρχές συμπεριλαμβανομένων και των δικαστηρίων και των δημοτικών συμβουλίων και αφορά και έγγραφα που κατέχουν ιδιώτες εφόσον χρησιμοποιούνται σε δημόσιες δραστηριότητες. Ο ορισμός του εγγράφου είναι ουδέτερος και καλύπτει μεγάλο φάσμα μηνυμάτων και εγγράφων που προετοιμάζει κάποια αρχή ή που υποβάλλονται σε κάποια αρχή. Όλα τα έγγραφα που μπαίνουν στο δημόσιο τομέα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν ενωρίτερα πρόσβαση σε όλους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει το δικαίωμα περιορισμού μόνον εάν δεν έχει ακόμη τελειώσει η διεκπαιρέωση και καταχώρηση ή εάν υπάρχει συγκεκριμένο συμφέρον για απαγόρευση. Οι δημόσιες αρχές επίσης έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν απρόσκοπτα το δικαίωμα στην πρόσβαση. Αυτό σημαίνει ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, καλύτερη διαχείριση της πληροφόρησης και ιδιαίτερα είναι υποχρεωμένες οι δημόσιες αρχές να πληροφορούν για το ποια έγγραφα κατέχουν ποια νομοσχέδια προετοιμάζονται και ποιες αποφάσεις προετοιμάζει η κυβέρνηση. Φυσικά το δικαίωμα πρόσβαση στα έγγραφα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα που πρέπει να προστατευτούν και γι' αυτό το νομοσχέδιο αυτό έχει και μακρύ κατάλογο εξαιρέσεων. Οι περιορισμοί εξαιρέσεις αυτές έχουν συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τη βασική αρχή της διαφάνειας και απαγορεύεται η πρόσβαση μόνον σε ό,τι θεωρείται απολύτως απαραίτητο να απαγορευτεί, δηλαδή ζωτικά ή επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντα ή θέματα διεθνούς συνεργασίας. Ακόμη πιο σημαντικό, οι περισσότερες εξαιρέσεις βασίζονται την αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και των συμφερόντων που μπορεί να βλάψει η δημοσιοποίηση. Αυτή η εξισορρόπηση των δύο δικαιωμάτων και η στενή ερμηνεία οδηγεί σε ένα σύστημα όπου πολύ λίγα έγγραφα απαγορεύονται. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. τα ναύλα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δικαιολογητικά τους είναι δημόσια και των βουλευτών και όλων των άλλων δημοσίων υπαλλήλων και δημοσιεύονται ελεύθερα. Αν ένας υπουργός και τα έξοδα παράστασης επίσης δημοσιεύονται, αν ένας υπουργός προσφέρει γεύματα κτλ. Η Τράπεζα της Φιλανδίας έχει σοφέρ για επίσημα αυτοκίνητα και πρέπει ο σοφέρ κάθε φορά να γράφει και να υποβάλει πού πήγε, πότε γύρισε κτλ. Και είναι και αυτό δημόσιο. Τρίτο παράδειγμα, ακόμη πιο σημαντικό, υπάρχει μία πρόταση για τη φορολογία όπου μπορεί κάποιος δημόσιος υπάλληλος για τον υπολογισμό κάποιου φόρου να πει ότι οι υπολογισμοί που έκανα δεν είναι δημόσιοι, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα, όχι είπε το δικαστήριο. Όλοι οι υπολογισμοί των φόρων είναι και αυτοί δημόσιοι και επίσημοι. Τέταρτον και τελευταίον, οι επιχορηγήσεις προς τους γεωργούς έχουν συζητηθεί στη Φιλανδία και επειδή είναι δημόσιες επιχορηγήσεις είναι και αυτές δημόσιες. Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια αξιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής με κάποιο επικριτικό πνεύμα, κριτικό πνεύμα. Για μας το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι η πρόταση μεγάλους αριθμός εγγράφων ε, να βγουν από το εύρος του κανονισμού 1049. Αυτή η τάση που παρατηρείται θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των δημοσίων εγγράφων που θα χορηγούνται. Αυτό μπορεί να δημιουργεί λιγότερη γραφειοκρατία, αλλά είναι υπερβολικά εύκολη λύση. Γιατί πολλά από αυτά τα έγγραφα θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν το κοινό και δεν θα υπάρχει πια πρόσβαση. Η εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων απαιτεί και κάποιο κόστος. Και αυτό ισχύει και για την πρόσβαση στα έγγραφα. Το κόστος αυτό όμως εξισορροπείται από την μεγαλύτερη αξιοπιστία που δημιουργείται. Τέλος κυρίες και κύριοι θα ήθελα να τονίσω το ρόλο του κλίματος, του διοικητικού κλίματος που καλλιεργείται. Γιατί η διαφάνεια δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Φοβάμαι ότι η πρόταση της Κομισιόν δείχνει ότι η γενικότερη στάση προς τη διαφάνεια είναι κάπως περιορισμένη. Και μπορεί κανείς να φανταστεί ότι αυτό ισχύει και γενικότερα στο διοικητικό κλίμα της Ένωσης. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κίμων Σάση, που αποδεικνύει και η δική σας τοποθέτηση ότι πολύ ωραία επιλέξαμε τα μέλη του πάνελ μας διότι σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως εκείνη που γνωρίζω καλύτερα τη δική μου, ε, είστε σε πολύ καλό δρόμο και πολύ καλές πρακτικές σας. Θα δώσω το λόγο τώρα στους βουλευτές. Πέντε αμιλητές έχω αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε να καλύψουμε την καθυστέρησή μας, ε, θα είμαι λίγο αυστηρός και θα σας επιβάλλω ένα τρίλεπτο στον καθένα σας. συνάδελφος από την Ισπανική Γερουσία, Αρκάδιο Ντίας, Τεχέρα. Τεχέρα. Ε, Συζητούσα με τον ε, Ιταλό συνάδελφο. Ε, σας ευχαριστώ και να σας καλωσορίσω κύριε Σάση. Ξέρετε ότι είχαμε βρεθεί και στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και στην ε, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην Διέτα είχατε έρθει και γνωριστήκαμε εκεί. Νομίζω Το ζήτημα δεν είναι να υπογραμμίσουμε το κατά πόσο ευεργετούμεθα όλοι. Δηλαδή αν είμαστε τόσο καλοί, ε, δίκαιοι και ευεργετούμενοι ή ευεργετούμε, τότε γιατί συζητούμε αυτό το θέμα στο δυναικές. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι λέμε και τι κάνουμε. Τι γίνεται με τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Αυτή η διαφορά μεταξύ του λέγειν και των ε, νομοθετικών αποφάσεων και της πράξης σχετίζεται με τον ηρωισμό που θα πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης. Δηλαδή πρέπει να διαθέσει χρόνο, να πάει από γραφείο σε γραφείο και στο τέλος να μπορεί να ρίξει μία ματιά σε ένα μικρό, σε ένα απόσπασμα από αυτό που θα ήθελε. Και επειδή μιλάμε, είμαστε στο 2009, μιλάμε για θετική προσέγγιση του θέματος. Ήρθα σε επαφή με έναν γερουσιαστή και έναν δικηγόρο εδώ και αυτό που έχει σημασία είναι η προσβασιμότητα στην πληροφορία. Δεν πρέπει να είναι ήρωας ο πολίτης για να έχει πρόσβαση στην πληροφορία, γιατί δυστυχώς πρέπει να είναι ο υπερήρωας. Τη στιγμή που έχουμε αυτό το, αυτή την φοβερή μηχανή, το διαδίκτυο, τότε γιατί ο άνθρωπος θα πρέπει να μεταβεί ο ίδιος, να μιλήσει με πολλούς και να πάρει επί χάρτου πληροφορίες. Γιατί να μην έχει πρόσβαση από το σπίτι του σε πραγματικό χρόνο, πληκτρολογώντας να έχει τα πολεοδομικά σχέδια, τα χωροταξικά σχέδια, γιατί δηλαδή δεν μπορεί να λάβει τις ε, πληροφορίες εκεί, γιατί ας πούμε του χορηγήθηκε μία άδεια σε εκείνον, σε άλλον όχι και ούτω καθεξής. Γιατί πρέπει κανείς να μεταβεί για πληροφορίες και δεν μπορεί να τις ε, βρει από το σπίτι του, να τις έχει από το σπίτι του. Όπως ε, είπανε και οι δύο εισηγητές, για να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα από το σπίτι θα πρέπει να προωθηθεί έτσι ώστε να μην είναι κανείς ήρωας για να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και να μπορεί να έχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο. Ωραία. Τρία λεπτά ακριβώς, αγαπητέ συνάδελφε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Τιερή Πονάνσκι. Πιέρι Πονάνσκι από την Βουλή των Αντιπροσώπων της ε, Τσεχίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το λόγο. Το προηγούμενο θέμα, καθώς και το τωρινό, εντάσσονται στα πλαίσια της διαφάνειας και της καλύτερης ε, ορατότητας. Νομίζω ότι η Επιτροπή το 2006 εκκίνησε με αυτή την πρωτοβουλία περί διαφάνειας. Μου έκαναν εντύπωση ορισμένα στατιστικά στοιχεία και θα ήθελα να σας τα αναφέρω διότι ελέγχθη ότι υπάρχουν 2.500 οργανώσεις λόμπι, 1.500 παρασκηνιακοί φορείς και 4.300 έχουν καταγραφεί, δηλαδή ε, ελέγχονται κατά κάποιο τρόπο. Οι παρασκηνιακές δραστηριότητες μπορούν να είναι χρήσιμες, τα λόμπι μπορεί να είναι χρήσιμα, να μας δώσουν ορισμένες ε, επαγγελματικές πτυχές ή ιδέες σε σχέση με την εφαρμογή έμπρακτα των μελλοντικών ε, νομοθετικών προτάσεων. Αλλά οι στατιστικές αυτές μας δείχνουν ότι η πλειοψηφία αυτών των δραστηριοτήτων λαμβάνουν χώρα χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε για έναν ορισμό των δραστηριοτήτων λόμπι δηλαδή δραστηριότητες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτός ο ορισμός μου δείχνει ότι αυτές οι παρασκηνιακές δραστηριότητες είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, καθώς και για τους βουλευτές, θα πρέπει να υπάρχει κάποια δυνατότητα περιορισμού αυτών των ε, επιθετικών δραστηριοτήτων. Διαφορετικά, οι πολιτικοί στην ουσία πλήττονται δυσανάλογα. Άρα δεν θα πρέπει να μιλάμε για αναθεώρηση αυτών των εγγράφων ως προς τις παρασκηνιακές δραστηριότητες και να μιλάμε για δεσμευτική καταχώρηση θα φτάσουμε σε μια σωστή εξισορρόπηση του τι είναι νόμιμο και τι όχι. Ποιες παρασκηνιακές δραστηριότητες δηλαδή είναι νόμιμες και ποιες όχι. Και οι καταχωρημένες ε, οργανώσει ή φορείς θα πρέπει να δέχονται έναν κώδικα δεοντολογίας και να έχουν και σαφή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πολάνσκι. Πράγματι θίγεται ένα πολύ σημαντικό σημείο ο κύριος Αντρές Γκαλασόφσκι από την ε, Πολωνική Βουλή. Έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι σε αυτό το πολικό ψύχος της Βορείου Ευρώπης κάτι θα πρέπει να υπάρχει γιατί έχουμε τα δύο αυτά σκανδιναβικά παραδείγματα, πολύ καλά παραδείγματα σε σχέση με την πρόσβαση στα έγγραφα και την διαφάνεια στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και άρα θα πρέπει να συγχαρώ τους Σκανδιναβούς. Στην Πολωνία οι πολίτες είναι πεπισμένοι ότι τα επίσημα έγγραφα δηλαδή αυτά που λαμβάνουν από το διαδίκτυο δεν είναι πλήρη έγγραφα. Γι' αυτό θεωρούν ότι θα πρέπει να αποτανθούν σε έναν υπάλληλο που δουλεύει στη δημόσια διοίκηση για να έχουν κάτι το πιο απτό, πιο συγκεκριμένο. Αυτή είναι η κληρονομιά μας από την εποχή του κομμουνισμού. Δηλαδή δεν λαμβάνουμε τα έγγραφα από το διαδίκτυο, απευθυνόμαστε σε έναν υπάλληλο για να δούμε, α, υπάρχουν χρήματα για τις κοινοτικέ επιδοτήσεις. Δηλαδή νομίζει ο πολίτης ότι θα λάβει κάτι περισσότερο διαζώσεις. Οι αλλαγές γίνονται πολύ αργά. Οι πολίτες δεν φταίνε πάντα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από το διαδίκτυο, αλλά δεν είναι πάντα οι πληροφορίες που απαιτούνται από τους πολίτες. Η υπουργό μας ανέφερε κάτι το συγκεκριμένο. Υπάρχουν και αρνητικές πρακτικές, ιδιαίτερα στην ε, Πολωνία. Υπάρχει το Ινστιτούτο Ιστορικής Μνήμης, το οποίο συλλέγει τα αρχεία των ε, πρώην μυστικών υπηρεσιών της ε, Πολωνίας, της εποχής του κομμουνισμού. Και θα ήθελα να τονίσω ότι οι επιστήμονες και οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Πολλές φορές υπάρχουν διαρροές, δηλαδή πληροφορίες που φτάνουν, μέχρι τους δημοσιογράφους, αλλά όχι όπως θα ήθελαν. Άρα πολλές φορές δεν υπάρχει επιρροή στην διαχείριση της πληροφορίας. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις εμπιστευτικές ε, πληροφορίες και στις ε, δημόσιες, δημοσιοποιημένες. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, κατηγορίες ανάμεσα στους πολίτες που έχουν ευκολότερη ή δυσκολότερη πρόσβαση στους πολίτες. Δηλαδή οι πληροφορίες είναι είτε δημόσιες είτε εμπιστευτικές. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκαλασόφσκι. Το λόγο ο Τζάκομο Σαντίνη από την Ιταλική Γερουσία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχει νόημα να διευρύνουμε τη συζήτηση για τη διαφάνεια στην οποία αναφερθήκαμε πριν ως προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά η αρχική όθηση για τον πολίτη δίνεται από τα εθνικά κοινοβούλια, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ευκολότερη και πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα, αλλά πρωταρχική πρόσβαση στην ε, προπαρασκευή των νόμων. Δηλαδή πριν ε, εφαρμοστεί ή τεθεί σε ισχύ ο νόμος. Αυτό γίνεται από ομάδες πίεσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την ΟΚΕ ή την Επιτροπή Περιφερειών που προβάλλουν ε, ένα θετικό λόμπινγκ. Εμείς επικρινόμαστε για πολλά πράγματα στην Ιταλία και σε αυτό το τομέα. Έχουμε ένα νόμο από το 1990 που ενέκρινε το Ιταλικό Κοινοβούλιο που αναφέρεται στη συμμετοχή του πολίτη στο διοικητικό γίγνεσθε. Από τότε που ετέθησε εφαρμογή αυτός ο νόμος, όλες οι πράξεις της δημόσιας διοίκησης, της κυβέρνησης, των, της Βουλής των Αντιπροσώπων της Γερουσίας, όλες οι πράξεις είναι στη διάθεση του πολίτη με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Δηλαδή για λόγους καθαρά ιδιωτικού χαρακτήρα, εμπιστευτικού και ούτω καθεξής. Ήδη στην Ιταλία χρησιμοποιούνται τεχνολογικά μέσα και οι συζητήσεις που γίνονται στο Κοινοβούλιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή στη Γερουσία ε, μεταδίδονται από το διαδίκτυο. 30 λεπτά μετά, δηλαδή γίνεται αναμετάδοση με διαφορά χρόνου 30 λεπτά. Και γίνονται και ειδικέ αναμεταδόσεις. Άρα φτάνουμε και σε μία απλούστευση των σχέσεων με τον πολίτη και το Κοινοβούλιο δεν έχει αυτή την επιπρόσθετη εργασία διότι ο πολίτης αν θέλει ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να συμμετέχει και στο γίγνεσθε της δημόσιας διοίκησης. Και έτσι παραπονείται λιγότερο ο πολίτης και υπάρχουν και λιγότερες προσφυγές κατά της ε, δημόσιας διοίκησης. Και εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε για την ευθύνη, την θεσμική μας ευθύνη. Δεν πρόκειται για μία μάχη μεταξύ πολίτη και δημόσιας διοίκησης. Είναι δικαίωμα του πολίτη για να αποκατασταθεί η αλήθεια ή μία βλάβη. Δηλαδή ε, πρόκειται για υποχρέωση του, της δημόσιας διοίκησης. Ο πρόεδρος μου λέει ότι πρέπει να τελειώνω και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι ο πολίτης θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα και να είναι σίγουρος ότι δεν θα υπάρχουν συνέπειες για αυτή τη δράση έναντι της δημόσιας διοίκησης και δικαιοσύνη, δικαίωμα της δικαιοσύνης και δίκαιες εφαρμογής σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ κύριε Σαντίνη. Θα δώσω τώρα το λόγο. Κλείνει το μικρόφωνο του Πρόεδρου δυστυχώς. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να συνεισφέρω πολύ σύντομα στη συζήτηση αυτή, αν μου επιτρέπετε. Συζήτηση για τη διαφάνεια για τι ευρωπαϊκέ νομοθετικέ διαδικασίε. Μιλώ εξ ονόματο τη τσεχική γερουσία, που παρακολουθεί πολύ στενά ε, όλε τι ευρωπαϊκέ ε, πρωτοβουλίε σχετικά με την καλύτερη νομοθεσία, τη βελτίωση λήψης αποφάσεων και των αντιστοίχων διαδικασιών. για θέματα διαφάνειας ε, κτλ. Η γερουσία μας μελέτησε όλες τις νέες διατάξεις που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας και ε, ε, στοχεύουν στην αύξηση της διαφάνειας και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια πρωτοβουλία που υποβλήθηκε στη ε, Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων της Ιερουσίας, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, και αφορά την καλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης των νομοθετικών αποφάσεων, στην προπαρασκευή των νόμων και τη δυνατότητα υποβολής λεγόμενων συλλογικών σχολείων. Τι είναι αυτά όμως τα συλλογικά σχόλια, collective comments. Υπάρχουν ορισμένοι πολίτες που έχουν συλλογικά αιτήματα και θα πρέπει να την χάνουν Αντίστοιχη και ίση μεταχείριση με όλους του υπόλοιπου ε, ενδιαφερόμενους που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη νομοθετικών αποφάσεων. Και θα πρέπει μάλιστα να είναι υποχρέωση ε, του νομοθέτη να ε, δημοσιεύει όλα τα έγγραφα και ακόμα και τα νομοσχέδια πριν ψηφιστούν. Δυστυχώς η πρόταση αυτή δεν ευδοκίμησε διότι δεν συμφώνησε το νομοθετικό σώμα της Βουλή δηλαδή. Ε, πάντως υπάρχουν ήδη υπουργεία που ε, δημοσιεύουν νομοσχέδια ε, ή προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου. Για παράδειγμα, πρόσφατα εγκρίθηκε ο νέος ποινικό κώδικας ή ο εργατικός κώδικας, όπου το αρμόδιο κάθε φορά Υπουργείο συγκέντρωσε πάνω από 10.000 σχόλια πολιτών κατά την νόμο Παρασκευή. Βεβαίω ε, αυτή η συμμετοχή θα πρέπει να είναι προτεραιότητα, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ τη συνάδελφό μας, Βιρίνα Ριπέροβα, και δίνω μέσα το λόγο στο Μαωρίσιο Τούρκο από τη Βουλή της Ιταλίας. Μαωρίσιο. του Συμβουλίου μας είπε ότι θα πρέπει πριν ε, να δημοσιοποιούνται τα έγγραφα να υφίστανται έναν έλεγχο περί ωφελήμου ή μη χαρακτήρα. Μην ξεχνάμε την απόφαση του ΔΕΚ όπου 13 δικαστές ομόφωνα καταδίκασαν το Συμβούλιο και πολιτικά και νομικά δηλαδή και το Συμβούλιο και τη Νομική Υπηρεσία και της Επιτροπής και του Συμβουλίου για έλλειψη διαφάνειας. Δηλαδή επειδή δεν θέλησαν να δώσουν έγγραφα, να κοινοποιήσουν έγγραφα μέσα στα πλαίσια μιας διοικητικής διαδικασίας. Τότε ήμουν βουλευτής όταν έκανα αυτή την καταγγελία και κατά συνέπεια την προσφυγή. Ε, κύριε. Υπουργέ, εκτιμώ ιδιαίτερα την παρέμβασή σας και ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια του ΔΕΚ, διότι το βασίλειο της Σουηδίας ήταν η μόνη παρεμβαίνουσα χώρα υπέρ ημών. Γιατί οι πολίτες μας θεωρούν ένα ιδιωτικό κλαμπ. Και δεν ότι έχω την εντύπωση, έχω τη σιγουριά γι' αυτό, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή, τι θα κάνει το βασίλειο της Σουηδίας έτσι ώστε να δημοσιοποιήσει τις αποφάσεις των εθνικών αντιπροσωπιών στα πλαίσια του Συμβουλίου τη στιγμή που δεν λαμβάνονται αποφάσεις ομόφωνα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ε, ε, Ευχαριστώ Μαουρίσιο. Εδώ έληξε ο κατάλογος των μιλητών, εκτός αν θέλει να ζητήσει κανείς το λόγο ή τον είχε ζητήσει και δεν είχαμε σημειώσει το όνομα. Όχι. Υποθέτω ότι μιλήσατε όλοι όσοι θέλατε. Θα δώσω τώρα το λόγο με την αντίστροφη σειρά στους εκπροσώπους ε, του πάνελ. Πρώτος ο κύριος Κίμος Σάση για να απαντήσει και στη συνέχεια η Υπουργός ε, Μπέατρης Άσκ. Σε σχέση με τις πληροφορίες μέσω διαδικτύου, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι αρχές να διαδίδουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο και να υπάρχει ελεύθερη και εύκολη ε, πρόσβαση. Όμως δεν έχει νόημα να διατίθενται όλες οι πληροφορίες στο διαδίκτυο, δηλαδή οι αποδείξεις εξόδων των ε, υπουργών. Εάν τις βάλουμε στο διαδίκτυο θα έχουμε σωρία πληροφοριών και δεν θα μπορέσουμε να διακρίνουμε τις ουσιώδεις από τις ε, πουσιώδεις. Είναι σημαντικές πληροφορίες, οι σημαντικές μάλλον μπαίνουν στο διαδίκτυο. Αν όμως ένας υπουργός συμπεριφέρεται κατά τρόπο ύποπτο, θα μπορεί κανείς να πάει στο Υπουργείο και να πει «Α, θέλω να δω τα δικαιολογητικά εξόδων ενός Υπουργού», εάν υπάρχει κάποια αμφιβολία. Εάν υπάρχουν δηλαδή αμφιβολίες, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης πρόσβαση, αλλά στο διαδίκτυο εντάσσουμε τις ε, πιο σημαντικές πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους πάντες. Βεβαίως, αν το διαδίκτυο είναι τόσο δύσχριστο που δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο κοινός πολίτης, τότε πάλι δεν υπάρχει διαφάνεια. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε απλά συστήματα για τους πολίτες τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιούν τη στιγμή που δεν ξέρουν τους νομικούς τίτλους για να ξέρουν ποιο ακριβώς κεφάλαιο θα πρέπει να ανοίξουν. Σε σχέση με τους κανόνες για τις ομάδες πίεσης, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες Δηλαδή οι κανόνες δεν είναι το πρόβλημα για την επικοινωνία, γιατί η επικοινωνία θα πρέπει να είναι δυνατή. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η διαφάνεια. Αν έχουμε επαφές ε, έτσι ώστε όλα να είναι δημόσια, ε, στοιχεία, οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση και τα εθνικά κοινοβούλια να μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση εάν υπάρχουν κενά να ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες από μια συγκεκριμένη πηγή. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Σε σχέση με τις διαρροές, αν ε, γνωρίσει κανείς, έχει γνώση που δεν έχει κανένας άλλος, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ως πολιτικό μέσον. Άρα με τη διαφάνεια απαγορεύεται αυτό η ιδέα της διαφάνειας σχετίζεται με το ότι ο καθένας έχει την ίδια γνώση, τις ίδιες πληροφορίες και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο γνώσης, έχει ίσους όρους πρόσβασης δηλαδή, για να μην ε, έχει μοναδική ή μεμονωμένη πρόσβαση στη γνώση. Αν υπάρχουν ε, διαρροές σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Και έτσι ακριβώς ε, λειτουργούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τη δεκαετία του 90. Δηλαδή υπήρχε διαρροή πληροφοριών προς συγκεκριμένες εφημερίδες για να προωθήσουμε ορισμένα ζητήματα. Δεν είναι ο σωστός τρόπος. Θα πρέπει να γίνεται εξισορροπημένη συζήτηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων για να έχουμε ένα πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα. Σε σχέση με τις εθνικές ε, θέσεις, και την ε, ε, δημοσιοποίηση τους πριν ε, λάβει τελικές αποφάσεις το Συμβούλιο. Εδώ είμαι ιδιαίτερα προσωπικά προσεκτικός. Ήμουνα υπουργό και είχαμε ζητήσει από το Κοινοβούλιο να υπάρξει μία ευελιξία. Βλέπουμε πολλές φορές πώς γίνονται γνωμοδοτήσεις στην Κόρεπερ πριν από τις συναντήσεις του Συμβουλίου και μπορεί να επέλθουν αλλαγές. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να δημιουργηθεί αυτό το περιθώριο ευελιξίας και να αλλάξει η θέση. Εάν έχουμε εκ των προτέρων ε, δημοσιοποιημένες θέσεις, είναι πολύ δυσκολότερο να είναι κανείς ευέλικτος. Άρα η λήψη αποφάσεων είναι πιο δύσκολη. Θα ήταν καλύτερα βεβαίως να δημοσιοποιούνται οι εθνικές θέσεις των εθνικών αντιπροσωπιών έτσι ώστε να ξέρετε ποια είναι η θέση της Φιλανδίας, άλλων αντιπροσωπιών και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε στην χώρα να γίνεται μια ουσιώδη συζήτηση επί του θέματος. Εκεί υπάρχουν διάφορες γνώμες και η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει μια συγκεφαλαίωση της συζήτησης και να ασχοληθεί με όλες τις θέσεις, δηλαδή να συντάξει όλες τις θέσεις. Εάν προσπαθούμε να λάβουμε αποφάσεις με 27 χώρες, ξέρετε ότι συρρυκνούται η ευελιξία και ε, σέβομαι την απόφαση των χωρών να μην δημοσιοποιούνται οι θέσεις τους πριν από την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών. Μετά όμως πρέπει να δημοσιοποιούνται. Ξέρουμε λοιπόν πώς άρχισε η διαδικασία, μετά την αναλύουμε, βλέπουμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και μπορεί κανείς να κρίνει την πολιτική διαδικασία, όπως και εμείς ακριβώς κάναμε. Και οι πολίτες μπορούν να μας επικρίνουν, αν το θέλουν. Δηλαδή, οι πολίτες να έχουν το δικαίωμα να σχολιάσουν την όλη διαδικασία κατόπιν της λήψης των αποφάσεων ή της απόφασης. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η Υπουργό ευχαριστω πολυ το λογο εχει η Μπεατρίς Άσκ, για να απαντήσει. Δεν θα απαντήσω όλα όσα ελέγχναν, γιατί νομίζω ότι πολλά απαντήθηκαν εκ των προτέρων. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς χρησιμοποιείται και το διαδίκτυο. Ε, όπως και στις περισσότερες χώρες και στη Σουηδία παρέχονται πολλές πληροφορίες. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Βεβαίως ε, δεν είναι πλήρης ε, οι πληροφορίες. Η δημόσια διοίκηση αποφασίζει ποιες πληροφορίες ε, διαβιβάζει, αλλά αυτό δεν επιλύει το πρόβλημα ως προς την ανάγκη Υπάρχουν πολλά διοικητικά προγράμματα όπου προσπαθούμε να εντάξουμε περισσότερες δραστηριότητες, να τις αναφέρουμε στο διαδίκτυο. Θα δούμε το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας και βεβαίως οι πολίτες μπορούν να έχουν τα έγγραφα μέσω email σήμερα αν το επιθυμούν. Αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι πολλά, τα, πολλά έγγραφα δεν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει αυτή η φόρμα και γι' αυτό δεν μπορούμε να τα εντάξουμε στο διαδικτύο. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μια καταχώρηση στο ίντερνετ έτσι ώστε να ξέρουν ε, οι πολίτες τι υπάρχει και έτσι έχουν ε, ευκολότερη πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες και μετά να τις ε, ζητήσουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει. Ο Πολωνός βουλευτής μίλησε για τις ομάδες πίεσης και τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά από την άλλη πλευρά η διαφάνεια αφορά το δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση. Το θέμα με τις ομάδες πίεσης πρέπει να το χειριστούμε διαφορετικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λανθασμένο μέσο προς μία κατεύθυνση που είναι σωστό σε μία άλλη. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η πρόσμιξη. Δεν έχει νόημα να σταματήσουμε τις ομάδες πίεσης κλείνοντας την πόρτα στους πολίτες το οποίο θα ισχύσει αν χρησιμοποιηθούν αυτοί οι κανόνες που ισχύουν για τις ομάδες ε, πίεσης. Ως προς τις διαρροές, συμφωνώ με τον Φιλανδό συνάδελφο και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι στην επόμενη Προεδρία θα λάβουμε τις πληροφορίες που θέλουμε από το ΔΕΚ και πέρα από τα προβλήματα που υπάρχουν διότι οι πολιτικοί μιλάνε, μιλάνε πολύ όταν θεωρούν ότι δεν έχουν στοιχεία την επόμενη μέρα. Εάν υπάρχει, υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να προωθήσουν τη θέση τους στα ΜΜΕ άμεσα το κάνουν. Αλλά χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα μετά τη Χάγη μακροχρόνια σε σχέση με τη διαφάνεια, την σαφήνεια, την σαφή γλώσσα. Και τώρα αναμένουμε την έκθεση της Επιτροπής το Μάιο και κατά τη Σουηδική Προεδρία θα εργαστούμε επί του προγράμματος και θα το εντάξω αυτό το πρόγραμμα στην εργασία μου. Δεν είναι εύκολο να εξευρεθούν κανόνες, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι να εργαστούμε με την Επιτροπή σε θέματα διαφάνειας, διότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία, στα τα οποία θα μπορούσαμε να χειριστούμε λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Όπως προβλέπετε θα δώσω τώρα το λόγο για να ε, ολοκληρώσει στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κύριο Νικηφόρο Διαμαντούρο, ο οποίος είναι πραγματικά ο κατάλληλο άνθρωπο γιατί παίρνει τα άπονα και τι καταγγελίε των πολιτών και έχει πραγματική εμπειρία ω προ την απογοήτευση των Ευρωπαίων πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανα και τι πολιτικέ τη. Του ζητήσαμε λοιπόν να διαπραγματευτεί το εξή θέμα. Με ποιο τρόπο, πώ μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευση για τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι βέλτιστε πρακτικέ των κρατών μελών σχετικά με τη διαφάνεια και την ορθή διακυβέρνηση. Νομίζω ότι ε, άκουσε με πολύ μεγάλη προσοχή τους δύο προλαλήσαντες. Κύριε Διαμεσολαβητά, έχετε το λόγο. Merci beaucoup, Monsieur Président. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα προσπαθήσω να αποφύγω τα προβλήματα της απογοήτευσης και να επικεντρωθώ στα προβλήματα της διαφάνειας και της ορθής διακυβέρνησης. Θα σας μιλήσω στα αγγλικά, μου επιτρέπετε, γιατί αγγλικά προετοιμάστηκε η ομιλία μου. Πριν πω στην προετοιμασμένη ομιλία μου, επιτρέψτε μου σύντομα να κάνω κάποια αυθόρμητα σχόλια. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Υπουργό κυρία Άσκ και τον κύριο Σάση τα όσα μας είπαν πάρα πολύ διαφωτιστικά και ενημερωτικά, όχι μόνο για μένα, γενικότερα για όλους. Και για μένα ως διαμεσολαβητή ήταν πολύ ενημερωτικά και διαφωτιστικά για ε, περαιτέρω ε, περισυλλογή και σκέψεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφάνεια, όχι μόνο για το διαμεσολαβητή, αλλά και για την ένωση ολόκληρη. Θα ήθελα εδώ να σας πω ότι προφανώς η διαφάνεια, η εμπιστοσύνη, η νομιμότητα, η λογοδοσία Ακόμα και η απλή ε, γλώσσα και η απλή διατύπωση είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπω και στο δικό μου θεσμικό όργανο, αλλά κανένα από όλα αυτά δεν είναι αυτοσκοπή. Είναι μέσα προς το στόχο και ο στόχος ουσιαστικά ποιος είναι ε, σε αυτή τη συγκεκριμένη ε, ιστορική συγκυρία, πώς θα φέρουμε την Ένωση καλύτερα, κοντύτερα στους πολίτες, πώς θα ενισχύσουμε τη δυνατότητα μεγαλύτερης εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τον κύριο Μαωρίσιο Τούρκο. Τούρκο διότι αποτελεί απόφαση σχετική Τούρκο ε, ε, στο 10 ορόσημο για το διαμεσολαβητή. Έχει ανοίξει νέες οδούς, νέες λεωφόρους για διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προσφυγή του στο ΔΕΚ και δικαιώθηκε. Και δικαιώθηκε και η θέση του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή πριν από 7 έτη. Ε, πρόεδρε, αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα όσο να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε να συμμετάσχω στην κοινή σας αυτή συνεδρίαση και που μου ζητήσετε να μιλήσω για το πώς μπορούν να εμπνευστούν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών σχετικά με τη διαφάνεια και την ορθή διακυβέρνηση. Σε μια δημοκρατία η διαφάνεια και η ορθή διακυβέρνηση σημαίνει να δίνουμε την ισχύ και την εξουσία στους πολίτες. Όπως φαίνεται από την αντίστοιχη σύμβαση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για την πρόσβαση στα έργα ε, σημαίνει καλή διακυβέρνηση η διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι εκείνη που επιτρέπει στους πολίτες να ασκούν έλεγχο ε, στις ε, δραστηριότητες των κρατικών αρχών, να αξιολογούν τις πρακτικές τους και να τους κάνουν να λογοδοτούν. Επίσης οι πολίτες μπορούν να ασκούν και τα άλλα τους πολιτικά δικαιώματα όπως η ελευθερία της έκφρασης και η συμμετοχή στα κοινά πώς μπορούν να εμπνευστούν καλύτερα από τα κράτη-μέλη και τις βέλτιστες πρακτικές. Το πρώτο έχει να κάνει με την νομοθετική διαδικασία. Εξ όσων γνωρίζω, Κανένας ε, δεν αφισβητεί σοβαρά ε, ότι η νομοθετική διαδικασία στα κράτη-μέλη είναι και θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανής. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε επίπεδο Ένωση. Δηλαδή τον Οκτώβριο του 2005 συνέστησα το Συμβούλιο να αναθεωρήσει την άρνηση του να ε, συνεδριάσει δημόσια όταν συνεδριάζει με την ομοθετική του ιδιότητα. Τον Απρίλιο του 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που υποστήριζε τη δική μου σύσταση. Ωστόσο, παρόλο που έχει γίνει κάποια πρόοδο σχετικά, το Συμβούλιο ανθίσταται και δεν ε, συμμορφούνται ακόμα πλήρω ε, προ τι υποδείξει και τις συστάσεις. Στα κράτη-μέλη ε, αυτό ε, δεν το διαπραγματεύονται τα κράτη-μέλη. Γιατί είναι δεδομένη η διαφάνεια στην νομοθετική διαδικασία και τώρα περνούν στο προπαρασκευαστικό στάδιο, αλλά στην Ευρώπη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει άσκηση πίεσης πριν ε, και μετά την εφαρμογή ε, δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συμπεράσματά της στη μελέτη αντικτύπου και λοιπά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η, λιμένη ε, απόφαση για την νομοθεσία. Επίσης υπάρχει ένα σύστημα μητρώου και καταγραφής των ομάδων πίεσης. Βεβαίως αυτό χωρίς καμιά αμφιβολία σημαίνει ένα βήμα προς τα εμπρός για τη διαφάνεια όσο και χωράει ακόμα βελτιώσεις. Βεβαίως η διαφάνεια του λόμπι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σε πολλά κράτη-μέλη σήμερα. Η διαδικασία αυτή, ο κανονισμός 1049 ε, του 2001 για τη διαφάνεια αφορά και ε, τη διοικητική εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εφαρμογή και επιβολή του Ευρωπαϊκού νόμου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ευρώπη δεν πρόκειται να έρθει πιο κοντά στους πολίτες απλώς εγκρίνοντας καλές ε, πολιτικές και καλούς νόμους. Εάν οι πολιτικές και οι νόμοι δεν εφαρμόζονται, δεν επιβάλλονται σωστά, τότε δεν θα έχουν κανένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Η διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη διοικητική εργασία, το σύνθες έργο, είναι ε, εξίσου σημαντική με την ομοθετική διαφάνεια. Η διοικητική εφαρμογή των ευρωπαϊκών ε, πολιτικών και των κοινοτικών νόμων δεν είναι απλώς θέμα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Το αντίθετο, κατά πρώτο λόγο, είναι ευθύνη των κρατών μελών. Τα κράτη, οι πολίτες μάλλον που θέλουν να δουν πώς εφαρμόζονται οι κοινοτικοί νόμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θα πρέπει έτσι να ψάξουν μέσα 28 ε, κανονισμούς και κανόνες, όχι μόνο το 1049, ε, που αφορά τα τρία θεσμικά όργανα, ε, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή, αλλά υπάρχουν από εκεί πέρα 27 ένομες τάξεις στα κράτη-μέλη. Και υπάρχουν και κάποια κράτη που έχουν και περιφερειακή νομοθεσία που έρχεται να περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές για ε, πρόσβαση τους πολίτες των μελών που θέλουν να ελέγξουν πόσο αποτελεσματικές είναι οι πολιτικές και οι της Ένωσης. Από την άλλη, Υπάρχει μια ποικιλία εθνικών νόμων που δίνει πολύ έδαφος για να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον, για να ε, αναλάσουμε εμπειρίες και πληροφορίες για τις βέλτιες πρακτικές. Ωστόσο, τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη δεν έχουν ένα βήμα για να συνεννοούνται για αυτά τα θέματα, για την πρόσβαση του κοινού σε κείμενα και έγγραφα και πληροφορία. Οι εθνικοί συνήγοροι του πολίτη, διαμεσολαβητέ, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, οι ομόλογοι μου με βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια να δούμε τι ισχύει στα διάφορα κράτη-μέλη και τι ε, τηρούν ως ε, στοιχεία τη τράπεζες δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα ε, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την πρόσβαση του κοινού γιατί είναι σωρία πραγματικά πληθώρα οι πληροφορίε που τηρούνται στα, στις βάσεις δεδομένων. Τώρα υπάρχει στη διάθεσή σας αυτή η μελέτη. Ελπίζω και πιστεύω να σας βοηθήσει να ενημερωθείτε για τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη-μέλη, αλλά και να βοηθήσει στη διάδοση αυτών των βέλτιστων πρακτικών. Πέρυσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, αναβάθμισε το καθεστώς μου, το ενημέρωσε καλύτερα ε, ως εθνικού ευρωπαϊκού διαμεσολαβητή, γιατί είμαι υποχρεωμένος να συνεργάζομαι όχι μόνο με τους συνηγόρους του πολίτη, τους εθνικούς, αλλά και με άλλες αρχές που πομίζονται την προστασία των ε, δικαιωμάτων και των δεδομένων. Εγώ ε, είμαι στη διάθεση σας να κάνω ό,τι μπορώ και ακόμα περισσότερα και να συνεργάζομαι με ε, εθνικούς αντίστοιχους ε, φορείς ε, πληροφόρησης και ε, αντίστοιχους παντού. Τέλος, θα ήθελα να διαπιστώσω με θλίψη ότι οι πολίτες αναλαμβάνουν την Ευρώπη ως ένα όργανο απόμακρο και μυστικό και ιδιωτικό. Με αυτό που θέλουμε εμείς να έχουμε κανόνες και στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη, αλλά με όσο γίνεται μεγαλύτερη πρόσβαση του κοινού. Για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες. Οι μόνοι που θέλουν ε, περιορισμό της πρόσβασης ε, των ε, πολιτών είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται να γίνονται μυστικές συμφωνίες και να αποφασίζονται στην Ευρώπη ορισμένα πράγματα μόνο από τους ηθήνοντες και κάποιες ομάδες πιέσεων και συμφερόντων. Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Δεν θα πρέπει μόνο τα θεσμικά όργανα αλλά και οι κρατικές αρχές να συνεργάζονται για να δημιουργηθεί μια τέτοια Ευρώπη ε, θα πρέπει οπωσδήποτε οποιαδήποτε αλλαγή στον κανονισμό 1049 του 2001 να είναι προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και μάλιστα ένα βήμα προς τη διαφάνεια και όχι ένα βήμα πίσω. Θα πρέπει πιο συστηματικά να ασχοληθεί η Ένωση πλέον με την πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα σε επίπεδο πλέον κρατών μελών για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, ε, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Διαμαντούρο για την εισήγηση αυτήν. Νομίζω όλοι κατάλαβαν το νόημά της. Ευχαριστώ επίσης την Σουηδέζα Υπουργό και όλους όσους παρενέβησαν και θα ζητήσω από τους δύο άλλους συμπροέδρους μας να έρθουν εδώ στο βήμα για να μας πούν τα συμπεράσματά τους. Και γνωστοποιώ σε όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων ότι το απόγευμα αν έχουν χρόνο και ενδιαφέρον η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών συνεδριάζει στις 3 και θα ακούσει τον κύριο Ζιλ Ντεκερκόφ που είναι ο Ευρωπαίος Συντονιστής για την καταπολέμηση της τρομοκαρατίας. Όσοι ενδιαφέρονται να ακούσουν τι μέτρα προβλέπουμε να ληφθούν μπορούν να προσέλθουν το απόγευμα στις 3 στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών γνωστή και ως ΛΙΜΠΕ. Υπάρχει συνέντευξη τύπου αμέσως μετά εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα την ίδια και πάλι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να την παρακολουθήσουν και τώρα επειδή ήρθε η ώρα των συμπερασμάτων Και επειδή εγώ είχα την τιμή να εγκαινιάσω την αρχή των ημερίδων θα δώσω το λόγο στους δύο συμπροέδρους για να μας εκφράσουν τα συμπεράσματα από τις συζητήσεις που είχαμε τις δύο αυτές, κατά τις δύο αυτές συνεδριάσεις. Ποιος θα αρχίσει πρώτος, ποιος... Ε? Υπάρχει ένας κανόνας ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προηγούνται οι γυναίκες. Γι' αυτό Πρώτα η κυρία Καπρικού, συμπρόεδρος, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέλεια. Καταρχάς, σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση τη χθεσινή και τη σημερινή. Διότι τέθηκαν πολλά θέματα και ερωτήματα και δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο από αυτά ως σημαντικότερο. Δεν έχω καμία προτίμηση. Αλλά ας συνοψίσω. Τη χθεσινή ίδιο συζήτηση, το βασικότερο νομίζω θέμα, το κρισιμότερο, και τήρηση της Οδηγίας 38 του 2004. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε πολλά και ακούσαμε πολλά διότι μάθαμε ότι όλα τα εθνικά κοινοβούλια αντιμετωπίζουν δυσκολίες με αυτή την οδηγία. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές διότι εξέφρασαν την προθυμία τους έτσι ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν διότι όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο για όλους. Και είμαι σίγουρη ότι θα φτάσουμε σε αυτό τον στόχο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να λειτουργήσει ε, σύμφωνα με αυτά τα νέα ε, δεδομένα και κανόνες. Θα ήθελα να μου πείτε όποτε έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε άλλα σοβαρά ε, ζητήματα και σας εύχομαι καλό ταξίδι στην ε, πατρίδα σας. Δίνω το λόγο τώρα στον δεύτερο συνπροεδρεύοντα, τον κύριο Σάτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και θα ήθελα να σχολιάσω τη συζήτηση που αφορά, αφορά την τρίτη συνεδρία. Στην τρίτη συνεδρία βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την αναθεώρηση του κανονισμού που αφορά την καλύτερη πρόσβαση σε, στην πληροφορία και έγινε και ένα σχόλιο ότι θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις όταν κάποιος αρνείται να παρέχει πληροφορίες. Και βεβαίως η αντίδραση που ακούσαμε ήταν ότι αν δώσουμε προτεραιότητα σε μια συγκεκριμένη ομάδα επαγγελματιών, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταχρήσεις. Και Η ομιλία της Επιτρόπου μας έδειξε ότι καταβάλλεται προσπάθεια βελτίωσης της διαφάνειας και ίσως η πρόταση του κανονισμού ε, δεν δείχνει αυτή τη θέληση τόσο σταθερά γιατί μιλάμε και για τον ορισμό των δημοσίων εγγράφων, τι θεωρείται δημόσιο έγγραφο και υπάρχει δυσκολία για την, ως προς την ε, πρόσβαση στην πληροφορία κατά την ε, προπαρασκευαστική νομοθετική διαδικασία. Άρα ίσως αυτή η αναθεώρηση να μην είναι η καλύτερη δυνατή. Δεν κινείται προς την ε, καλύτερη κατεύθυνση, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ότι ο κανονισμός ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ είναι αρκετά καλός και ιδιαίτερα χρήσιμος. Χάρηκα που άκουσα την Αντιπρόεδρο να μιλήσει για τα αποτελέσματα μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου και αυτό ε, αφορά και τα σχόλια του αναπληρωτή Υπουργού. Ξέρετε ότι η Επιτροπή δεν έχει και πολύ χρόνο στη διάθεσή της για αυτή την αναθεώρηση, αλλά δεν θα ήταν και σκόπιμο να επιταχύνουμε ιδιαίτερα αυτή τη διαδικασία, διότι αυτό θα έπλητε την σωστή πρόσβαση, καλή πρόσβαση στις πληροφορίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεπρέ, τον πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και τους άλλους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι δέχτηκαν την πρόσκλησή μας να συμμετάσχουν και χαίρομαι διότι είχαμε αθρώα προσέλευση με πολλά σχόλια και ελπίζω ότι αυτή η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών κοινοβουλίων θα είναι το καλύτερο παράδειγμα των πραγματικών μας αναγκών έτσι ώστε να μειώσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα στις νομοθετικές μας εργασίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ κύριε Ζεύτσικ. Το μόνο που απομένει είναι να σας πω εγώ μερικά συμπερασματικά. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Τσεχική Δημοκρατία για τη συνδιοργάνωση και συ-επιτυχία, θα έλεγα της κοινή αυτής ε, συνεδρίασης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εθνικών ε, Κοινοβουλίων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και όλους σας ανεξάρτητα από τις χώρες και τη Βουλή από την οποία προέρχεστε ή το κοινοβουλευτικό σας σώμα. Ε, πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά που μας είπατε. Συμπερασματικά νομίζω μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε στο εξή. Όλοι συμφωνούμε έτσι δεν είναι ότι ήταν παράλογο και άφρον να προσπαθήσουμε να χτίσουμε την Ευρώπη αντιμέτωπη και εις βάρος των κρατών. Μα ποτέ δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Τα κράτη συνεργαζόμενα οικοδομούν την Ευρώπη. Αντίστοιχα παράλογο θα ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεωρεί ότι μπορεί να νομοθετεί εις βάρος και απέναντι στους ε, εθνικούς νομοθέτες. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πόλεμος των νομοθετικών σωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και έχουν νόημα τέτοιες συνεδριάσεις και παρακαλώ πιστέψτε μας όταν σας λέμε ότι έχουν ουσιαστική σημασία για μας τέτοιου είδους συνεδριάσεις. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να γνωρίζουμε την άποψη των εθνικών κοινοβουλίων. Έτσι, γενικά και αόριστα. Επιζητούμε τη συνεργασία με τα κράτη μέλη. Διότι σε εμάς αναπόκειται να νομοθετούμε, αλλά ε, θα πρέπει να παίρνουμε και την άποψη εκείνων που ζουν στα κράτη-μέλη για να μην κάνουμε λάθη στις προτάσεις σας και στα όσα αποφασίζουμε για τα κράτη-μέλη και τα καλούμε να τα εφαρμόσουν. Και επίσης θέλουμε και συνεργασία στη μεταφορά. Γιατί εάν η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν ε, μεταφέρεται σωστά στα διάφορα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια χήμερα και πλάνη. Δεν έχουμε ε, νομική ε, συνάφεια και κάποια στιγμή θα εκτεθούμε και στα μάτια και ε, της κοινή γνώμης και των πολιτών μας. Δηλαδή πραγματικά θέλω να υμνήσω τη συνεργασία και την επιζητούμε και να μην θεωρούν ότι στα θεσμικά όργανα υπάρχει ε, αυτή η μυστικότητα το Αν μη τι άλλο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε να είμαστε πλήρως ε, ανοιχτοί, διαφανείς και να διαβιβάζουμε όλες τις προφορίες και να υπάρχει πάντα πρόσβαση στα έγγραφα. Και θα θέλαμε να είμαστε υπόδειγμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δώσουμε το καλό παράδειγμα για τις βέλτιστες πρακτικές που στο μέλλον θα ε, διευρυνθούν και θα εδραιωθούν. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και κηρύσω το πέρας της συνεδρίασης.